Varmt välkomna till eh, dagens möte Ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας για τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουμε μια ιδιαίτερα πεφορτωμένη ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό σας ζητώ να ξεκινήσουμε εγκαίρως. Πρώτο θέμα είναι η έγκριση μέσης διάταξης. Έχετε εδώ κάποιες παρατηρήσεις. Έχουμε μετά την έκθεση της κυρίας Οβίερ. την οποία θα την μετακινήσουμε την γνωμοδότηση της κυρίας Οβίερ. Δεν θα την εξετάσουμε το πρωί σήμερα. Αν λοιπόν συμφωνείτε με αυτή την αλλαγή για την ημέρα συνένταξη μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχετε από τη δική σας πλευρά για την ημέρα συνένταξη παρατήρησης Εξ της ε, ομάδας των φιλελευθέρων εγώ θα ήθελα να λάβω το λόγο να προσθεθεί αυτό το θέμα στην μέση διάταξη. Συγκεκριμένα, Θέλω να, να διαμαρτυρηθώ για την κατάρριση του, της, του Ρουμανικού Φορέα για την ισότητα των ε, φύλων. Μαζί με τον Φορέα για την Προστασία των Οικογενειών και των Παιδιών και τον Φορέα για την Προστασία των Αναπήρων καταργήθηκε στη Ρουμανία. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να καταργηθούν αυτοί οι φορείς γιατί αυτό συνεπάγεται έλλειψη σεβασμού για μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ισότητα ανδρών και γυναικών, και αυτό έγινε αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα όπου όλοι μας συμφωνήσαμε ότι δεν είναι παραδεκτό το να μην σεβόμαστε τα δικαιώματα <clears throat> και την ισότητα των φίλων λόγω της οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πληροφορήσω και να ζητήσω να καταγραφεί στα πρακτικά η διαματήρια μας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία που μας δώσατε. Μπορώ να σας πω και εγώ ότι έχω αποστείλει ήδη μια επιστολή που περιέχει αυτά τα οποία είπατε κι εσείς. και αυτή η επιστολή θα σταλεί και στους, εισηγη... στους συντονιστές μας. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της συνάντησης των συντονιστών σήμερα το απόγευμα στις 5.30 να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρατε. Μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι έχει γίνει δεκτή η ημερησία διάταξη για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ούτε έχει αφαιρεστεί, περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο να σας αναφέρω και περνάω κατευθείαν στο σημείο 3. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους μας και εμένα προσωπικά που εξ ονόματος της Επιτροπής μας μπορώ να καλωσορίσω τον Ζωζέ Μέντες Μπότα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Ισότητα Ευκαιριών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μέντες Μπότα υπήρξε στο παρελθόν Ευρωβουλευτής από το 1989 μέχρι το 1994 και στη συνέχεια από το 1998 στο 1999 και έχει συμβάλει σημαντικά στις εργασίες της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης και επίσης και της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Εμείς συναντιόμεθα σήμερα με τον κύριο Μπότα, ώστε να μπορέσει, να μπορέσει να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ της δικής μας Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε την κατάσταση των ίσων ευκαιριών σε όλη την Ευρώπη και της ισότητας των φίλων στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Μπότα, ώστε να μας παρουσιάσει <clears throat> την εργασία που εκτιλήσεται στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχετε το λόγο κύριε Μπότα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Με μεγάλη μου χαρά λαμβάνω το λόγο επί θεμάτων ίσης εκπροσώπης ανδρών και γυναικών στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου είμαι πρόεδρος από τον Ιανουάριο. Χαίρομαι που μπορώ να σας μιλήσω σε αυτούς τους καιρούς ε, μεγάλων αλλαγών. Ο ε, Γενικός ε, Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης και η κυρία Βίβιαν Ρέντιν, ε, Επίτροπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησαν για την συμμετοχή, μάλλον την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και δείξαμε θέματα νομικών προκλήσεων για το σύστημα, σημαντικό σύστημα της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως πρώην Ευρωβουλευτής, όπως σας υπενθύμησε και η Πρόεδρος, θεωρώ ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας παρέχει νέες ευκαιρίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Και έτσι μπορούμε να συνδράμουμε και οι δύο. Όπως θα τονίσω, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση προετοιμάζει μια έκθεση για τις επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας στο Συμβουλίο της Ευρώπης, που θα καλύψει αρκετές πτυχές ως προς τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης μετά την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας. Η ισότητα των δύο φύλων είναι ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος επιδιώκουμε τους ίδιους στόχους έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν περισσότερα δικαιώματα, να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη, ισότητα και περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες. Ελπίζουμε αυτή η στόχη να είναι συμπληρωματική. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε ορισμένα βασικά σημεία που βρίσκονται και στις ε, δύο ατζέντε μας έτσι ώστε να φτάσουμε σε εκπλήρωση στόχων με βάση τις κοινέ προσπάθειες. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την, το, εμπόριο ανθρώπων έτσι ώστε στα πλαίσια μιας μελλοντικής οδηγίας για την καταπολέμηση ε, εμπορίου ανθρώπων θα πρέπει να υπενθυμίσω το Συμβούλιο της Ευρώπησης μέσα στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας. Αυτή η οδηγία ε, ίσχυσε από την 1η Δευτέρου 2008 και 25 χώρες ε, έχουν κυρώσει αυτή τη σύμβαση, ενώ 15 άλλες έχουν κυρώσει και την οδηγία. Αυτό σημαίνει αφορά ε, χώρες διαμετακόμισης και χώρες υποδοχής και προορισμού. Όταν κυρωθεί η συνθήκη, τα κράτη θα συμβαδίζουν με ευρωπαϊκά πρότυπα και θα υπάρχει ένας εποπτικός μηχανισμός που ονομάζεται Γκρέτα. Η Γκρέτα, αυτός ο εποπτικός μηχανισμός, θα λογοδοτεί στις εθνικές αρχές. Είναι ένα δεσμευτικό όργανο. Αυτός ο ανεξάρτητος εποπτικός οργανισμός απαρτίζεται από 13 πρόσωπα, έτσι ώστε να εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτός εποπτείας για να αξιολογηθούν οι χώρες Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση εξέφρασε την ανησυχία της για την επικάλυψη εργασιών και τον ε, πολλαπλασιασμό κυρωτικών διαδικασιών και εποπτικών αρχών. Η κυρία Γιζέλα Βέρμ μίλησε για έναν παράγοντα κόποση που ίσως γνωρίσουν τα κράτη-μέλη στη διαδικασία αυτής της εποπτείας. Θεωρούμε ότι αυτή η επικάλυψη είναι δαπανηρή και θα, μπορούσε να, θα μπορούσαν να μην είναι σε θέση να την αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Η κυρία Λίδη Χέρ που συμμετέχει στην υποεπιτροπή ε, αυτή συμμετείχε σε ένα κοινό σεμινάριο για την κατάργηση της εμπορίας αυτής από τον Ιούνιο του 2010 και τόνισε ότι ο τρόπος εποπτείας είναι ίσω ίσως είναι διαφορετικό στη μελλοντική οδηγία με βάση τον ε, μηχανισμό εποπτείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ενθάρρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη Σύμβαση το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε τα ίδια, ίδιες προδιαγραφές να ισχύουν παντού δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πρότυπα αυτά του Συμβουλίου της Ευρώπης να είναι σημείο αναφοράς για όλα τα διεθνή μέσα και μηχανισμούς. Τα πρότυπα αυτά που θα καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μελλοντική της οδηγία θα πρέπει να είναι σύμβατα και εξίσου απαιτητικά με αυτά του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπ' αυτή την έννοια χαίρομαι διότι προωθείται ένας επικοδομητικός διάλογος με την πρόεδρο της Υποεπιτροπής ως προς το δουλεμπόριο και θα πρέπει να, ε, ε, να γίνει πιο εντατικός αυτός ο διάλογος κατά τους επόμενους μήνες. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμηθεί το δουλεμπόριο και γι' αυτό η Κοινοβουλευτική Συνέλευση θα ε, οργανώσει μια διεθνή διάσκεψη κατά του δουλεμπορίου στις 3 Δεκεμβρίου του 2010. Προσωπικά εξέφρασα στην Πρόεδρο την θέλησή μας να να συμμετάσχετε και θα θέλαμε και οι κοινοί οι της Επιτροπής σας και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ενισχυτικά. Καλό και τα μέλη αυτής της Επιτροπής να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διάσκεψη που θα οργανωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Στόχος είναι να λάβουμε υπόψη τη διεθνή εργασία μέχρι τούδε, τους ε, νομικούς μηχανισμούς, τους δεσμευτικούς μηχανισμούς, καθώς και την εργασία των ε, εθνικών κοινοβουλίων και όσων συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Θα ήθελα οι συνεισηγητές να συμμετάσχουν αν μπορούν. Τέλος, θα ήθελα να πω προς όλα τα μέλη της Επιτροπής ότι ε, έκανα μία υπόδειξη στην πρόεδρό σας από πλευράς Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για δύο τροπολογίες σε σχέση με την οδηγία επί του θέματος αυτού που θα σας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες και ιδιαίτερα τη δική σας Επιτροπή. Ως προς το άρθρο 13, η πρώτη τροπολογία αποτελεί παράδειγμα όπου θα θέλαμε να ε, διαιωνιστούν αυτά τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα θύματα δουλεμπορίου που δεν, έχουν, που δεν τους διέπει ένα νομικό καθεστώς ως προς τον τόπο διαμονής, αλλά που θα πρέπει να τύχουν αρρωγής όποτε χρειάζεται τουλάχιστον για μία περίοδο 30 ημερών που εξετάζεται ο φάκελός τους. Θα ήθελα να πω ότι αρχικά το Συμβούλιο είχε ασχοληθεί με το πρώτο προσχέδιο αυτής της οδηγίας. Δεν υπάρχει αυτή η αρχική περίοδος ε, περισυλλογής των 30 ημερών πλέον. Θα ήθελα να το σκεφτείτε έτσι ώστε να αρκεστείτε στα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά μία περίοδο περισυλλογής 30 ημερών. Ως προς το άρθρο 19.2 και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα αποφυγής επικάλυψης εργασιών και ενεχόμενου κόστους. Έχουμε ε, τη δική μας Επιτροπή Εποπτείας ως προς τη σύμβαση καταπολέμησης του δουλεμπορίου και εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, ε, παραγράφου, τότε θα προσθεθούν δύο επιπροσθέτως μηχανισμοί και αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε σε τρεις συνολικά μηχανισμούς και άρα τα κράτη θα γνωρίσουν αυτό το παράγοντα κόπωσης από την εποπτεία. Γιατί θα πρέπει να διερευνηθεί το όλο ζήτημα τρεις φορές για την καταπολέμηση δουλεμπορίου. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε την επικάλυψη δις και τρεις. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω αφορά την βία κατά των γυναικών. Και ε, εδώ θα πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα. Αυτή τη στιγμή συγγράφουμε μία σύμβαση για να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών και στα νοικοκυριά. Μέχρι το τέλος του 2010 θα πρέπει να καταρτιστεί το έγγραφο έτσι ώστε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης να μπορέσει να αποφασίσει μέσα στο 2011. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε απαιτητικέ προδιαγραφές σε σχέση με την αντιμετώπιση των θυμάτων και την δίωξη των θητών. Πιστεύω ότι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ισπανικής Προεδρίας και οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενίσχυση των μέτρων για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών, οι προτάσεις αυτές είναι πρόσδεκτες, διότι πρόκειται για κοινέ ε, προσπάθειες που καταβάλουμε για να μην δεχτούμε πλέον τη βία κατά των γυναικών. Έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πραγματικής ισότητας των δύο φύλων Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη των μέσων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση παρακολουθεί την εργασία μιας επιτροπής η οποία ε, συστάθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρατηρητής. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε τρεις νέες εκθέσεις μέσα στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας. Uh, uh, Και θα ήθελα να συνεργαστείτε επί των θεμάτων αυτών. Αντιμετωπίζουμε ε, ε, συγκεκριμένες προσφυγές για την αντιμετώπιση της βίας και βεβαίως θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την πορνογραφία και ιδιαίτερα την παιδική πορνογραφία για να την εντάξουμε στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Να υπάρχει λοιπόν προστασία των θυμάτων με βάση τη βία που βασίζεται στο φύλλο και το ε, Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να λάβει υπόψη και την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας με βάση την εφαρμογή και παρακολούθηση και έλεγχο της μελλοντική σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα ήθελα η Κομισιόν το συντομότερο δυνατόν να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ισομερή συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην λήψη αποφάσεων. Η κοινοβουλευτική συνέλευση θεωρεί ότι θα πρέπει να καταπονομήσει τη βία κατά των γυναικών μέσα στα πλαίσια της ίσης κατανομής εξουσιών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών έτσι ώστε να αλλάξουμε αυτό το, το πρότυπο συμπεριφοράς που υπάρχει και οι γυναίκες να βρουν τη θέση που τους αξίζει στις δημοκρατίες μας. Θα πρέπει λοιπόν να μην θεωρήσουμε ότι επιτελείται οπωσδήποτε πρόοδος ε, εκεί που δεν επιτελείται. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στη, στον πολιτικό βίο μέσω των εκλογικών συστημάτων και μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Είμαστε πεπισμένοι ότι αν δεν αλλάξουμε το εκλογικό σύστημα, εάν δεν υπάρχει έστω και προσωρινή προσωρινός υποχρεωτικός χαρακτήρας, τότε τα αποτελέσματα δεν θα είναι παρά απειροελάχιστα. Και θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, όπως τη Σουηδία που γνωρίζει, έχει μάλλον ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο. Έχω προωθήσει ε, διάλογο με χώρες της Λατινικής και Νότιας Αφρικής και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα ποσοστώσεων και εκεί ακριβώς εκπροσωπούνται περισσότερο οι γυναίκες στην κυβέρνηση. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα και γι' αυτό ε, πέρσι ε, δημιουργήσαμε αυτό το βραβείο για την ε, ισότητα μεταξύ των δύο φίλων και το οποίο απονείμαμε πέρσι στην σοσιαλιστική πολιτική ομάδα της Πορτογαλίας ε, για να δείξουμε με αυτό το γραφείο ότι ε, θα πρέπει πράγματι να διασφαλιστεί ότι έχουν πρόσβαση στις ε, θέσει των ερωτών εκπροσώπων οι γυναίκε μέσα στις πολιτικές ομάδες. Πολύ συχνά τα κόμματα κατηγορούνται για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημοκρατία ως καθεστώ, αλλά αποτελούν βασικού πυλώνε του δημοκρατικού συστήματο τα πολιτικά κόμματα και για παράδειγμα και μέσω αυτού του βραβείου μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα πολιτικά κόμματα εκείνα τα οποία έχουν προβεί και στις εξωτερικές και στις εσωτερικές εκείνες δράσεις που διασφαλίζουν να ε, κλέγονται περισσότερες γυναίκες να βραβεύονται για αυτά. Άρα λοιπόν θα ήθελα να βασιστώ και στη δική σας ε, συμβόλη ε, είτε είναι στα Εθνικά Κοινοβούλια, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε σε διεθνείς οργανώσεις. Μιλάμε δηλαδή για, κάτι, για μια ανοιχτή διαδικασία οποιοδήποτε δηλαδή μπορεί να είναι υποψήφιος ε, για το βραβείο αυτό. Η συνέλευση επίσης ασχολήθηκε το 2010 με την οικονομική κατάσταση των ε, γυναικών. Ε, αναφέρθηκε σε μία έκθεση σε ό,τι αφορά την διαφορά, τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φίλων, το ζήτημα των δίκαιων συντάξεων για τις γυναίκες και το Σεπτέμβριο στο Παρίσι θα οργανώσουμε μία ακρόαση ε, σε ό,τι αφορά την περισσότερη συμμετοχή των ε, γυναικών στις, ε, στα θεσμικά όργανα που είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων, γιατί πραγματικά θα θέλαμε να δούμε τις γυναίκες να λαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο σε κάθε είδους φορείς είναι για παράδειγμα πολύ σπάνιο το να δούμε μια γυναίκα να βρίσκεται επικεφαλής ενός αθλητικού ομίλου ή να βλέπουμε μια γυναίκα Βρίτανη είναι κάπως πάνω αυτό, τουλάχιστον σε κάποιε χώρες που γνωρίζω εγώ. Μα ανησυχεί λοιπόν αυτό. Επίση, ε, το ζήτημα των ε, ε, γυναικών στις αγροτικέ περιοχές είναι ένα ακόμα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε το 2011. Πριν επίσης ασχοληθήκαμε με την καταπολέμηση των σεξιστικών στερεοτύπων και πράγματι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις ε, ε, γυναίκες ε, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να υπάρχει μια εμπορική μεταχείριση αν θέλετε και να συνεχίζονται στερεότυπα τα οποία ίσιαν εδώ και χιλιετίες. Επίση, συζητούμε ένα νέο πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο ε, θα ε, διασφάλισε το θεμελιώδε δικαίωμα τη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και η δική μα ε, Επιτροπή για τι Ευκαιρίε ασχολήθηκε με μια έκθεση με αυτό το σημαντικό ζήτημα το οποίο θα οδηγούσε σε μια σημαντική αλλαγή των τρόπων με τον οποίο καταπολεμούμε τις να άνηση μεταχείριση μεταξύ των δύο όφελων. Ε, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρώ πω σε αυτή την περίοδο αλλαγών μα δίνονται νέε ευκαιρίε, νέε δυνατότητε για να κάνουμε και εμεί αλλαγέ. και νομίζω πω ε, έχουμε την πρόκληση απέναντί μα να ανεβάσουμε κι άλλο τον πύχη σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων και νομίζω πω μπορούμε να βασιστούμε στη δική σα επιτροπή ώστε να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ε, γυναικών ε, στην Ευρώπη και να προωθηθούν αυτά τα ζητήματα όχι μόνο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά ε, και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια των 27 κρατών Και επαναλαμβάνω ε, την πρόσκλησή μου στην οργάνωσή μα ε, στην εκδήλωση που θα έχουμε το Δεκέμβριο και αναμένω με ενδιαφέρον τι δικέ σα απόψει, τα δικά σα σχόλια ω προ το πώ μπορούμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η κυρία πρόεδρο. για την παρουσίασή σας, την οποία ακολουθήσαμε, παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρούμε ότι πράγματι στους δύο διαφορετικούς αυτούς χώρους στους οποίους εργαζόμαστε μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια συνεργασία προς τον κοινό σκοπό της υποστήριξης ισότητας των φύλων. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή σας να επισκεφθούμε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εμείς έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά που απασχολούν και τη δική σας επιτροπή, δηλαδή το λαθρεμπόριο ανθρώπων. Μας έχετε προσκαλέσει να επισκεφθούμε την επιτροπή σας το Σεπτέμβριο και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Μπορώ να ανοίξω τώρα τη συζήτηση. Η κυρία Μπάουερ έχει καταρχήν το λόγο. Έχετε το λόγο κυρία Μπάουερ. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ευκαιρία αυτή να έχω ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπότα και πιστεύω ότι αυτό είναι ένας πολύ τρόπος να προχωρήσουμε γιατί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβουλίο της Ευρώπης που είναι γείτονες πολλές φορές στο Στρασβούργο Εργαζόμαστε για τα ίδια θέματα πολλές φορές. Και πιστεύω ότι και αυτή είναι μια ευκαιρία που μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε, διότι μας απασχολούν τα ίδια προβλήματα. Και ένα από αυτά τα προβλήματα είναι το λαθρεμπόριο ανθρώπων, που συζητήθηκε και στην κοινή μας ε, συνάντηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για τις παρατηρήσεις σας σε σχέση με, την, τον χρόνο προβληματισμού. Εμείς έχουμε άλλο ένα νομικό εργαλείο, έχουμε προσωρινές άδειε διαμονής που καλύπτουν τα προβλήματα αυτά. Αλλά όταν δεν υπάρχουν αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να αναπληρωθούν Να διορθωθεί η κατάσταση λοιπόν των πολλών αυτών θυμάτων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προερχόνται από διαφορετικά κράτη-μέλη και θα πρέπει να καλύπτονται όλες αυτές οι δυνατότητες. Για την παρακολούθηση επίσης και την εποπτεία και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μας γιατί βασιζόμαστε στην περίπτωση αυτή σε δύο διαφορετικά νομικά εργαλεία. Η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι το ένα εργαλείο και αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς είναι ένα άλλο εργαλείο. Καλύπτουν διαφορετικές περιστάσεις βέβαια, αλλά επειδή υπάρχει μια κοινή προβληματική, μια κοινή θεματολογία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην, επικαλυφ... να μην επικαλύπτονται οι προσπάθειές μας, <clears throat> όπως είπατε, να μην υπάρξει κόποση παρακολούθησης για τα θέματα αυτά γιατί αυτό θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ούτως ή άλλως αντιμετωπίσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα με το υψηλό επίπεδο ανοχής που υπάρχει για τις περιπτώσεις ε, ε, λαθρεμπορίας ανθρωπίνων όντων, πολλά από τα οποία, πολλές από τις οποίες στην περίπτωση αυτή βρίσκονται και σε συνθήκες αναγκαστικής εργασίας καταναγκασμού να εργαστούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία στους τομείς αυτούς. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν Και φυσικά εδώ είναι και ένα θέμα χρόνου. Θα καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε Δεν ξέρω αν τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας θα μας δώσουν κάποια συγκεκριμένη διάταξη που να, επιτύχει την, να εξασφαλίσει την επιτυχία της συνεργασίας μεταξύ μας, αλλά βλέπω να υπάρχουν και προβλήματα βέβαια. Αλλά υπάρχει πραγματικά και η διαφορά προσέγγιση από τα δύο μας όργανα. Εμείς προσβλέπουμε με την ευκαιρία μιας, της νέας αυτής σύμβασης που αναφέρατε για τα προβλήματα αυτά αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα πιο αποτελεσματικά. και φυσικά όλα τα θέματα τα οποία αναφέρατε βρίσκονται σε άινα η συζήτηση μέσα στην Επιτροπή μας. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εγώ θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη μιας πιο στενής και υποφελούς συνεργασίας μεταξύ της δικής μας Επιτροπής και της Επιτροπής Συμβουλίου της Ευρώπης. Πιστεύω ότι η συνεργασία αυτού του είδους μεταξύ των δύο αντιστοίχων επιτροπών θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμη και εποφέλης αμοιβαία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος, κυρία Μπάουερ. Τέσσερις ακόμα ομιλήτριες στον κατάλογό μου. Θα πρότεινα να ομαδοποιήσουμε τις παρεμβάσεις αυτές και στη συνέχεια θα ξαναδώσω πάλι το λόγο στον κύριο Μέντις Μπότα για να μπορέσει να δώσει μια απάντηση. Η κυρία Στρέλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Μέντες Μπότα, παλιογνώριμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερος για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει στον τομέα της ισότητας των φύλων, για τον αγώνα του κατά όλων των μορφών διακρίσεως, ιδίω της βίας κατά των γυναικών και το λαθρεμπόριο λευκής σαρκός. Και θα ήθελα επομένω και πάλι να χαιρετήσω τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. <clears throat> Όλα τα θέματα τα οποία ανέφερε πράγματι είναι τμήμα και του δικού μας ενδιαφέροντος και των δικών μας ενασχολήσεων αναφέρθηκε σε μία σειρά από προτεραιότητες, από θέματα που μας απασχολούν σε επίπεδο προτεραιότητας και φυσικά οικοθενοείται ότι ο θεσμικός διάλογος μεταξύ των δύο οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πιο στενή συνεργασία είναι απόλυτα επιθυμητή και εποφελής εξάλλου. Και θα ήθελα τώρα να κάνω παρατηρήσεις σε σχέση με τα ζητήματα τα οποία ανέφερε ο κ. Μέντου Μπότα. Για το λαθρεμπόριο ανθρωπίνων όντων και ιδίως γυναικών και παιδιών, που είναι τα κύρια θύματα αυτής της λαθρεμπορίας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και πρόκειται κυρίως για γυναίκες οι οποίες υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση βρίσκονται σε μια νέα μορφή δουλείας, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν οι εθνικές νομοθεσίες, να υπάρξουν πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη και επίσης να υπάρξουν και πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλύτερη προστασία των γυναικών αυτών, γιατί όσο δεν υπάρχει νομοθετική προστασία για αυτές τις γυναίκες οι οποίες χρήζουν επίσης και ψυχολογικής υποστήριξης δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να στρέψουμε τις προσπάθειές μας εναντίον των εγκληματιών αυτών που είναι λαθρέμποροι ανθρωπίνων όντων αφενός και αφετέρου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερη προστασία και ψυχολογική υποστήριξη προς τα θύματα. Επίσης ό,τι αφορά την ε, βία που βασίζεται <clears throat> στο φύλλο. Ξέρουμε ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο πολλές γυναίκες στην Ευρώπη ως θύματα της οικιακής βίας. <clears throat> Όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Μεντεσπότα, η Ισπανική Προεδρία έδωσε μια μεγάλη όθηση στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Ήταν μια από τις προτεραιότητες που είχε τονίσει η Ισπανική Προεδρία και περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την προσπάθεια, την περαιτέρω όθηση που έδωσε η Ισπανική Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Βία κτλ. Ακόμα δύο παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτον να υπάρξει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι προφανές ότι οι γυναίκες θα πρέπει να βρίσκονται σε επίπεδο απόλυτης ισοτιμίας με τους άνδρες και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο και εδώ τίθεται και το θέμα της συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή προσωπική ζωή. Και κάτι το οποίο συνδέεται με το θέμα αυτό είναι και η ανα... με την ανάγκη συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων είναι και το θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στην λήψη οικονομικού χαρακτήρα αποφάσεων. Αυτό συνδέεται με τη γενική κρίση στα οικονομικά θέματα που έχει θίξει τις φτωχότερες οικογένειες και ιδιαίτερα τις γυναίκες <clears throat> και είναι γνωστό ότι οι γυναίκες δεν είναι αυτές οι οποίες μπορούν να επομιστούν την ευθύνη αυτής της κρίσης ούτε μία γυναίκα δεν είναι διοικήτρια κεντρικής τράπεζας στα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη απουσία των γυναικών από τις ε, θέσεις υψηλής ευθύνης στον οικονομικό στίβο. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όπως υπάρχει το σύστημα ποσοστώσεως για την εκπροσώπηση των γυναικών σε πολιτικό επίπεδο, θα πρέπει ένα παρόμοιο σύστημα να ισχύει για τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική λήψη αποφάσεων στις δημόσιες επιχειρήσεις ή στις ε, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείε, όπως έχει αποφασιστεί στην Νορβηγία από την εκεί συντηρητική κυβέρνηση. Ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν ποσοστώσεων, το οποίο μπορεί να δώσει θετικά αποτελέσματα για μια καλύτερη προστασία των γυναικών στον πολιτικό χώρο, το ίδιο σύστημα θα μπορούσε να επεκταθεί και στον οικονομικό χώρο και φυσικά <clears throat> αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα της διαφοράς αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το 2004 ήταν 15% κατά μέσο όρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τώρα η ψαλίδα έχει ανοίξει και η διαφορά είναι 18% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για, θα είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί η ισότητα λοιπόν των γυναικών και να εξασφαλιστεί ότι συμμετέχουν στην αγορά εργασίας σε ποιήσεις όρες. Ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Στρέλα. Η κυρία Μπάστος, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ε, χαιρετήσω το συνάδελφο ο οποίος ε, ακολούθησε πολιτική σταδιοδρομία, τον κύριο Μέντες Μπότα και χαίρομαι που τον βλέπω τώρα ως εκπρόσωπο μιας επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες σε σχέση με την πολύ θετική εργασία, με το πέρασμα των χρόνων και τη συμμετοχή, ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ζούμε σε μία κοινωνία η οποία ολοένα και εξελίσσεται και γι' αυτό επαναπροσδιορίζουμε τις προτεραιότητές μας διεξοδικά όπως είπε και ο κύριος Μέντες Μπότα, για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, ιδιαίτερα της βίας σε επίπεδο νοικοκυριών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη συμμετοχή των γυναικών στην δημόσια ζωή, στην πολιτική ζωή. Σε αυτή την ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή και, συμμετοχή και το πώς συμβαδίζει με την οικογενειακή ζωή. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα, ιδιαίτερα στην κοινωνία μας που ζει μία μεγάλη κρίση αξιών Άρα η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας. Θα πρέπει να υπάρχει ίσιμη, ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, όπως ε, ισχύει για τους άνδρες. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Θα πρέπει να μπορούν να ακολουθήσουν μια πολιτική σταδιοδρομία ή γενικότερα επαγγελματική σταδιοδρομία, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να συνδυάσουν αυτή τη ζωή με την οικογενειακή ζωή. Ένα άλλο ζήτημα σχετίζεται με την κρίση που ζούμε, γιατί οι γυναίκες είναι τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της κρίσης με επιπτώσεις ε, επιπτώσεις στην ζωή, στον εργασιακό τομέα. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι γυναίκες κατέχουν διαφορετική θέση στην αγορά εργασίας, άρα είναι πολύ πιο εύκολο να απολυθούν. Πρόκειται για μια κατάσταση που οθεί τις γυναίκες προς την φτώχεια. Ένα άλλο ζήτημα έχει σχέση με κοινωνικές ανισορροπίες που οδηγούν σε ρήξη της οικογενειακής ζωής, ζωής ή περιθωριοποιεί τις γυναίκες και τις οθεί στην πορνεία ενδεχομένως. Είναι μια κατάσταση για την οποία θα πρέπει να εξεύρουμε απαντήσεις και ιδιαίτερα να ε, βρούμε δυναμικά μέτρα για την ε, αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων. Επίσης, ένα άλλο θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ σχετίζεται με την εργασία, με τις εργασίες στην Επιτροπή Κρίσης και τον επιχειρηματικό κόσμο όπως εξελίσσεται με τη συμμετοχή των γυναικών. Θα πρέπει οι γυναίκες να είναι αυτάρκεις ως ε, προς την πρόσβαση στην εργασία. Το επιχειρηματικό πνεύμα θα πρέπει να διακρίνει και τις γυναίκες, να μπορέσουν να συμμετέχουν στον επιχειρηματικό κόσμο και να ε, δημιουργούν ΜΜΕ, όπως οι άνδρες. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η θέση σας σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπάστος. Συγκλέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλώς ήρθατε, κυρία Μπότα. Στο συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ προηγουμένω κατά τη δική σα παρουσίαση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έγινε για, το, την εμπορία ανθρώπων, που αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε πως η Συμφωνία να αποτελεί πρόβλημα ε, για αυτό το θέμα. Ε, δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι, ε, έχουν τη δυνατότητα ε, οι άνθρωποι να μετακινούνται, να περνάνε πάρα πολλά σύνορα χωρίς ελέγχους, άρα ίσως οι διάφοροι δουλεύουν είναι σε σε θέση να ε, ε, προβαίνουν σε αυτέ τι δραστηριότητε. Μήπω θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι στα σύνορα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική ζωή, εγώ να σας πω πως ε, ε ευρωβουλευτής χωρίς ε, να χρειαστεί να υπάρξει κάποια θετική διάκριση υπέρ μου και είχα και μία συνάδελφο που είχε ε, κάνει ακριβώ το ίδιο για πάρα πολύ καιρό με, με δική μας ε, πρωθυπουργό. Μετά είχαμε μία κυβέρνηση των εργατικών που είχε αυξηθεί εκεί το ποσοστό των γυναικών με μία σχετική ποσόστοση και από, έως το 2002 υπήρχε ήδη ένα σημαντικός αριθμός γυναικών και από εκεί και μετά δεν ενδιαφέρονταν πλέον ε, ενδεχομένως οι γυναίκες ή ε, για παράδειγμα δεν συμμετείχαν καν στις εκλογές και να θυμίσω ότι το 1997 ε, είχαμε κάποιες εκλογές όπου είχε γίνει μία βασική αλλαγή και εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι πως σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε τους καλύτερου υποψήφιου για μια συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή, διάκριση όποια και αν είναι δεν μπορεί να είναι θετική, α το πούμε έτσι. Δηλαδή η δική σα χάρτα είναι μια χάρτα υπέρ τη διακρίση κατά κάποιο τρόπο. Άρα είμαι κατά αυτή τη χάρτα. Επίση, λέτε πω ε, δεν υπάρχουν για παράδειγμα οι ε, ε, σε ποδοσφαιρικού οπλού που είναι γυναίκε. Αλλά από το Birmingham, τα West Midlands, έχουμε την κυρία Μπρίντ που είναι η... είναι πράγματι επικεφαλή εκεί ενός αθλητικού Άρα λοιπόν θα ήθελα να συμφωνήσω και με την προηγούμενη ομιλήτρια. Δηλαδή το ζήτημα εδώ, το πρόβλημα είναι η οικογενειακή ζωή και οι υποχρεώσεις της, ε, όχι ε, το φύλλο. Δηλαδή να προβλέψουμε ότι υπάρχουν ε, τα, οι, οι σωστές υποδομές σε ό,τι αφορά την ε, περίθαλψη, την φροντίδα για τα παιδιά, τη δυνατότητα δηλαδή να, να λάβουν κάποια εργασία οι γυναίκες. Έτσι μπορούμε να έχουμε σωστή μεταχείριση και όχι το αντίστροφο. Uh, Να χαιρετήσω τον πρώην συνάδελφό μας, τον κύριο Μέντες Πότα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι είσαστε ιδιαίτερα αφοσιωμένος στο έργο σας ως πρόεδρος της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και επίσης χαιρετίζω ιδιαίτερα τη συμμετοχή σας, όπως και πολλών άλλων ανδρών, στις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της οικογενειακής βίας που στρέφεται κατά των γυναικών. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε πείσει ακόμα και περισσότερους άνδρες κοινοβουλευτικού να συμμετέχουν σε τέτοιες επιτροπές, γιατί όταν μιλάμε στους άνδρες για τα θέματα αυτά, γελούν μαζί μας. Επομένως, συμμερίζομαι απόλυτα όλες τις ανησυχίες που έχετε αναφέρει στη συζήτησή σας σήμερα το πρωί, στην παρουσίασή σας διότι το Συμβούλιο της Ευρώπης όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινού στόχους, έχουν παρόμοιους στόχους και ο κύριος, η κύρια αποστολή της Επιτροπής μας εδώ είναι να δώσουμε ίδια, ίσα δικαιώματα στις γυναίκες και να εξαλείψουμε κάθε μορφή διάκρισης εναντίον των γυναικών που να οφείλεται στην ε, λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων, την βία εναντίον τους, την ελλειπή συμμετοχή τους. Ελπίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε και ξέρω ότι υπάρχουν και επίσημες, σε επίσημο επίπεδο επαφές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο <clears throat> είναι απόρρια της, έγκριση της ε, έγκρισης της συνθήκης της Ευρώπης και θα ήθελα να ξέρω και ποια είναι η θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τις πρόνοιες αυτής της ε, συνθήκης γιατί ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτού που γίνεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό είναι απαραίτητο να μην υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση, αλλά ούτε και περί τι επικάλυψης της προσπάθειας μας. Επίσης, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε και περισσότερα άτομα να εργάζονται προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων παρά την καλή θέληση που υπάρχει, έχουμε μακρό δρόμο να διατρέξουμε στον τομέα αυτό. Και τέλο θέλω να τονίσω ότι είναι κεφαλαιώδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει και να ενσωματώσει όλα τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης ό,τι αφορά στην λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων, την έννοια της ε, προστασίας, της πρόληψης αλλά και της δίωξης των ενόχων. Υπάρχουν αυτά τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρέπει να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει, να προσχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στη σύμβαση για την προστασία των ε, θυμάτων λαθρεμπορίου κτλ. και να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζονται αυτά τα πρότυπα σε όλη την Ευρώπη με ομοιόμορφο τρόπο και θα είναι τα σημεία αναφορά για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλέ φορέ διαφορέ και ποικιλίε σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων, ακόμα και μεταξύ χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε ένα κοινό σημείο αναφορά, μια κοινή στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τη λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων. Σα ευχαριστώ πολύ και σα καλωσορίζω και πάλι. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρο. Η κυρία Χιμένεθ. Καλημέρα σας. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ κύριε Μεντεσπότα. Και θα σας έλεγα ότι δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο με όλα αυτά που είπατε και ήταν μια μεγάλη χαρά να ακούσω την δική σας άποψη γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία όπως ξέρετε μας απασχολούν και εμάς που συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που λέτε. Αναφέρθηκε πάρα πολύ το θέμα της βίας κατά των γυναικών και έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα να σας θέσω εδώ σε σχέση με αυτό διότι Είμαι η συγγήτρια μιας έκθεσης, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας των Θυμάτων σε τέτοιου είδους ε, πράξεις βίας και έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει την προστασία των θυμάτων, αλλά είναι λογικό ότι εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην προστασία των γυναικών που είναι πολλές φορές θύματα βίας λόγω φύλου. είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια που καταβάλουμε να υπάρξει μια αναμόρφωση και βελτίωση της νομοθεσίας για τα θέματα αυτά στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Θεωρείτε ότι θα είναι εύκολο να εφαρμοστεί μια τέτοια νομοθεσία ή θα έχουμε προβλήματα στην εφαρμογή. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό. Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Χθες είχα βρεθεί σε μία συνδιάσκεψη όπου μία δικηγόρος και ακτιβίστρια συγχρόνως αναφέρθηκε στα θέματα των γυναικών στο Ιράν και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά κυρίω στη δική της χώρα στο Ιράν. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο επίση έλαβε χώρα μια ακρόαση για τα προβλήματα πολλών νέων κοριτσιών στην Ευρώπη που ζουν ουσιαστικά σε καθεστώς δουλεία στην οικογένειά τους και πολλές φορές δολοφονούνται από την ίδια την οικογένειά τους γιατί επιλέγουν να ζουν σαν Ευρωπαίες μέσα σε εισαγωγικά. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία και εμείς στην Επιτροπή μας έχουμε την υποχρέωση να το εξάρουμε το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα και ποια είναι η αντιμετώπιση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Κύριος έχει και πάλι το λόγο για να απαντήσει στα ερωτήματα που σας ευχαριστώ πολύ όλους ε, για τα ενδιαφέροντα σχόλια που κάνατε και τα ερωτήματα που θέσατε. Θα προσπαθήσω να περιορίσω την παρέμβασή μου στα 5 λεπτά που μου αναλογούν για να προσπαθήσω να απαντήσω στα κυρία θέματα. Ε, στην κυρία Μπάουερ θα έλεγα το εξή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο μερικέ ε, φορέ να προβένουμε σε αυτή την ευαισθητοποίηση. Έχουμε δύο, δύο διαφορετικά εργαλεία. Αλλά ας το αποφύγουμε. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας, στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα σύστημα για την ε, ενημέρωση για την υποβολή εκθέσεων και δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η αλληλεπικάλυψη με τι αρμοδιότητε, δηλαδή με τα όσα κάνουμε και εμεί από την πλευρά του Συμβουλίου τη Ευρώπη. και ταυτόχρονα και τα κράτη-μέλη ε, κάνουν το ίδιο. Δηλαδή, ένα κράτο μέλο, είναι μέλος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλο του Συμβουλίου τη ε, Ευρώπη, και κατά συνέπεια καλείται επανειλημμένα να συντάξει τρει διαφορετικέ εκθέσει, οι δύο διαφορετικέ εκθέσεις για το ίδιο ακριβώ ζήτημα. Άρα λοιπόν, αν μπορούσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των τριών εκθέσεων σε δύο ή σε μία, θα ήταν κάτι το θετικό. Και συμφωνώ και με τα όσα είπατε, κυρία Παρόν σε σχέση με την συνεργασία. Τώρα να μιλήσω πορτοκαλικά. Σε σχέση με την αγαπητή κυρία Εστρέλα, συμπατριώτησα, θα ήθελα να της πω ότι καταλαβαίνω ότι πολλές χώρες αντιμετωπίζουν διαφορετικές καταστάσεις. Υπάρχουν χώρες που έχουν προηγμένη νομοθεσία και άλλες όχι. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία σύμβαση που είναι ένα δεσμευτικό κείμενο για τις ε, χώρες που το κυρώνουν που την κυρώνουν και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τους δουλεμπόρους και να προστατεύσουμε τα θύματα. Διότι σε αυτό το τομέα νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Υπάρχουν πολλά θύματα που φοβούνται να καταγγείλουν παρόμοιες καταστάσεις και υπάρχουν και απειλές κατά των οικογενειών τους. Γι' αυτό έχουμε να κάνουμε με ένα ε, κρυφό φαινόμενο, δηλαδή ένα φαινόμενο εγκρυπτό. Υπάρχουν απειλές, πιέσεις, εκβιασμοί κατά των οικογενειών, γι' αυτό τα ε, θύματα δέχονται αυτή την ε, κατάσταση, την απαράδεκτη κατάσταση. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε τις αστυνομικές έρευνες για να αποκαλύψουμε αυτά τα φαινόμενα και να κινηθούμε πέρα από την άκρη του παγόβουνου. Δηλαδή, με βάση αυτή την ζήτηση ε, που υπάρχει, κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες και τη στιγμή που ε, παρέχεται και προωθείται η πορνεία κατά τέτοιον απροκάλυπτο τρόπο, πίσω από όλες αυτές τις αγγελίες υπάρχουν οργανωμένοι, υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα και οργανωμένα δίκτυα που ε, υποχρεώνουν τις γυναίκες να εκπορνευτούν κατά τη θέλησή τους. Γι' αυτό έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η σύμβαση. Εμείς δεν θέλουμε πια άλλα κείμενα που να αποτελούν νεκρό γράμμα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί παρακολούθησης που είναι ύψης της σημασίας. Θα πρέπει να είναι πολύ ε, καλοί αυτοί οι μηχανισμοί και να προβλέπουν μια ευρύτατη εποπτεία. Αυτός είναι και ο ρόλος του κοινοβουλευτισμού, των εθνικών κοινοβουλίων, του ευρωπαϊκού. Υπάρχουν και παγκόσμιες οργανώσεις, διότι εμείς είμαστε ο κρίκος μεταξύ του κοινοβουλευτισμού και των πολιτών. Εμείς έχουμε εκλεγεί άμεσα από τους πολίτες Γι' αυτό ακριβώς στα πλαίσια αυτής της σύμβασης κατά της βίας που πλήττει τις γυναίκες και ιδιαίτερα και στον ιδιωτικό βίο, θα πρέπει ένας μηχανισμός εποπτείας να έχει μία κοινοβουλευτική προσέγγιση, δηλαδή οι βουλευτές να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία εθνικά. Επίσης, θα πρέπει να συμφιλειωθεί η επαγγελματική και η οικογενειακή ζωή. Και γι' αυτό χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι δεν έχει κανένα νόημα να προετοιμαζόμαστε από πολιτικής πλευράς αν δεν δημιουργήσουμε και τις κατάλληλες συνθήκες συμβατότητας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Θεωρούμε ότι είναι ένα βασικό θέμα ανησυχίας και γενικότερου μελήματος η χρηματοπιστωτική κρίση βεβαίως πλήττει πρωτίστως τις γυναίκες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, διότι στην ανεργία προωθούνται πρώτα οι γυναίκες, οι χαμηλόμιστες είναι οι γυναίκες και παρά την κρατική στήριξη, η κρατική στήριξη δόθηκε προς τομείς όπου δεν έχουν προεξάρχοντα ρόλο οι γυναίκες. Αυτοκινητοβιομηχανία, η μεγάλη πλειοψηφία που εργάζεται εκεί είναι οι άνδρες. Χρηματοπιστωτικός ε, τομέας. Ποιος ελέγχει αυτό το τομέα, οι άνδρες. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Γιατί στον τομέα της τραπεζικής αυτοκρατορίας δεν υπάρχουν γυναίκες. Η Φιλανδία διενέργησε μία μελέτη που καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις όπου προεξάρχοντα ρόλο παίζουν οι γυναίκες είναι ε, αυτές όπου συνδράμουν, και, συνδράμουν οι γυναίκες. Και αυτό αφορά και τα εμπορικά επιμελητήρια, όπως μας είπε και η κυρία Γκοτιέ. Τώρα, εντάχει, θα επεκταθώ και σε κάτι άλλο. Για την κυρία Ρεζίνα Μπάστος θα ήθελα να πω ότι η κρίση έχει και μία άλλη συνέπεια. Εγώ πίστευα ότι η βία στα νοικοκυριά ήταν ένα ε, θέμα που ήταν σταθερό. Απλώς οι καταγγελίες ήταν περισσότερες. Δηλαδή οι γυναίκες ευαισθητοποιήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Αυτό πίστευα ένα χρόνο πριν. Δυστυχώς όμως αυξάνεται η ιδιωτική βία. Κυρία Σίνκλερ, λυπάμαι διότι δεν συμμερίζομαι την άποψή σας. Διαφωνώ πλήρως. Ναι, υπάρχουν γυναίκες δηλαδή που έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει θετική διάκριση προς όφελος τους, αλλά δυστυχώς αυτές οι γυναίκες αποτελούσαν εξαιρέσεις Γενικά δηλαδή τα ποσοστά των γυναικών σε πολλά από αυτά τα θεσμικά όργανα δεν θα είναι δυνατόν να αυξηθούν χωρί να ληφθούν κάποια περισσότερα μέτρα. Ναι, κύριε Παπαδοπούλου, ναι, συμφωνούμε. Είναι δύσκολο δηλαδή να αντιμετωπίσουμε του άντρε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Ε, Κάθε χώρα είναι διαφορετική και στο Ιράν οι γυναίκε έχουν μεγάλε δυσκολίε να εκφραστούν, να ζήσουν ω Ευρωπαίε όπως και στις δικές μας χώρες πολλές φορές οι γυναίκες που έρχονται από ισλαμικό πλαίσιο έχουν δυσκολία να ε, συμπεριφερθούν ως Ευρωπαίες και είναι υποχρεωμένες να δίνονται με τον Ισλαμικό τρόπο. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει για λόγους <clears throat> θρησκευτικού ή άλλους να απαγορεύεται η χρήση της μπουρκας ή άλλων Ισλαμικών ενδυμάτων, αλλά για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που να περιορίζουν αυτή τη χρήση. Ευχαριστώ πολύ. Εξ τη Επιτροπής μας θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Μέντσου Μπότα για την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πολύ καλή συνεργασία που έχει υπάρξει μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. Ευχαριστώ. Και τώρα. Ερχόμαστε στην ε, ψηφοφορία. Σας παρακαλώ να πάρετε τις κάρτες ψηφοφορία σας και ερχόμαστε στην έκθεση της κυρίας Πιέτη Κάινεν στο ρόλο των γυναικών σε μια γυδάσκουσα κοινωνία και το ρόλο των γυναικών στη σύνολη κοινωνία όχι μοναχά των γυναικών βέβαια έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο, αλλά είναι ιδιαίτερος και ο ρόλος των γυναικών. Η κυρία Πίτικα είναι, είναι η συντάκτρια αυτής της ε, έκθεσης και θα να δώσω λόγο στην κυρία Πίτικα είναι για μια σύντομη παρουσίαση. Και σας παρακαλώ, σιωπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για την πολύ καλή συνεργασία τους σε σχέση με την έκθεση αυτή και για τις πολλές πολλές τροπολογίες οι οποίες βελτιώνουν την έκθεση. Έχουμε και μία συμβαστική τροπολογία η οποία συμπυκνώνει πολλές προτάσεις ιδίως σε ό,τι αφορά τις ασθένειες οι οποίες είναι ιδιαίτερες για τις γυναίκες Και σας υπενθυμίζω ότι η τροπολογία 67 δεν έχει ακόμα, δεν έχει πράγματι αποσυρθεί μεν, αλλά βρίσκεται, καλύπτεται πια από την ε, από την παγιοποιημένη τροπολογία συμβέσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία τι Ψηφίζουμε τώρα. Τροπολογία 15, ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απέριπτε 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, άποχες, δεκτό το πρώτο τμήμα. 2 υπέρ. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, μάλιστα. Το πρώτο τμήμα της 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφία. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται she didn't she didn't mention it before, so but I think we can we can vote Okay, we have voted and uh, Ψήφισαμε και απεριφθεί. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της 21. Ψήφι υπέρ του δεύτερου τμήματος 21 κατά αποχές. Δεκτό το δεύτερο τμήμα. Πάλι έλεγχο θέλετε. Καλά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία έλεγχο. The vote is η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό 14 Τροπολογία 22 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α, 20 την πηδήξαμε. Τώρα πάμε στην 22. Ψήφι υπέρ 22. Έλεγχος για την 22 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 22 που σας είπα προηγουμένως. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 25 έχει εκπέσει 26 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Έλεγχος για την 27 δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 28. Παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά, υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος για το 44 τμήμα 2 άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed and it's adopted. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ Α, καταπίπτει, με συγχωρείτε. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. 50 τμήμα δεύτερο. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is Πέρας. Απορρίπτεται λοιπόν. Τρίτο τμήμα της 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. 50 τμήμα τρίτο. Αρχίζει η ψηφοφορία. The Πέρας. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 56 α, καταπίπτει 30 υπέρ. Όχι, όχι, την διορθώνουν την πρόεδρο. Με συγχωρείτε, κανένα λάθος, λέει η Πρόεδρος. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Α, καταπίπτει, με συγχωρείτε. 61. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 65. 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η 77 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, ακαταπίπτει με συγχωρείτε. 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 82. Ωραία, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 81 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. Και η 86 λέει πρόεδρος 85. Με συγχωρείτε, έχω κάποιο πρόβλημα με τα έγγραφά μου. 87. 85. we have to vote on 85. Ψηφίζουμε την 85 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 87. 86 έξι. Υπέρ. 86 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 87. Θέλετε να ελέγξουμε την 86. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 86. Πέρας. Απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, α όχι πίπτη, λέει η πρόεδρος, 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες. Συμφωνείτε? Ψηφίζουμε από κοινού. Από την 9 μέχρι τέλους. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία επί του κειμένου και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά. Να συγχαρούμε την κυρία Πίτι Κέινεν, την εισηγήτρια. Nu går vi till eh, nästa ärende som också är en omröstning. Τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Είναι η έκθεση Bauer. Είναι έκθεση για γνωμοδότηση. Η Επιτροπή Απασχόλησης είναι η Επιτροπή επί της ουσίας. Δίνω το λόγο στην κυρία Μπάουερ. Εάν έχει παρατηρήσεις πριν από την ψηφοφορία. Έχετε το λόγο κυρία Μπάουερ. Δεν έχω και πολλά να πω. Να πω. Έχω την εντύπωση ότι σε μερικές ε, περιπτώσεις οι τροπολογίες αποτελούν βελτίωση και σε άλλες όχι. Μου φαίνεται όμως ότι ε, ίσως αποτελούν ε, βελτίωση στην έκθεση Thomas Mann. Ε, Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Ωραία, περνάμε στην ψηφοφορία τώρα. Υπέρ της 10 κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται 12 σε τέσσερα τμήματα, 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 15 σε δύο τμήματα. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16. Θέλετε να ελέγξουμε την 15, το δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία επί του δευτέρου τμήματος. Πέρας και απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 με μία προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. 22 δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει. Τρία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 4 καταπίπτει. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οκτώ υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και θέλετε να ελέγξουμε ωραία αρχίζει η ψηφοφορία πέρας και απορρίπτεται απορρίπτεται ένα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και να συγχαρούμε την κυρία Μπάουερ. Francisco Mai. Okay. So, I understand that everybody's... Από ό,τι καταλαβαίνω, όλοι ε, είναι μετά την ψηφοφορία κάπως έτσι σε μια πορεία δυναμική. Στις 2 ε, Ιουλίου η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων ε, Εθνών ε, προέβη στην ε, υιοθέτηση ενό ψηφίσματο που μα ενδιαφέρει και ε, νομίζω πω θα έπρεπε να τους αποστείλουμε μια συγχαρητήρια επιστολή για να το για να, το, για να εκφράσουμε τη δική μας συμπαράσταση. Θα το κάνουμε μέσω της δικής μας αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη. Και σε ό,τι αφορά ε, την αναφορά που μας έκανε η συνάδελφος ε, σε ό,τι αφορά την αρχή για την ε, ισότητα μεταξύ των δύο φίλων, δηλαδή κατάσταση τη Σχετική Επιτροπή στη Ρουμανία, να αποστείλουμε και για αυτό το ζήτημα μία επιστολή στη Ρουμανία. Δεν μπορεί δηλαδή λόγω μια οικονομική κρίση να γίνονται περικοπέ και απλά να καταργείται ένα θεσμό όπω αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σα κάνω αυτή τη σύσταση να αποστείλετε αυτέ τι δύο επιστολέ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νταμάη σε ό,τι αφορά το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, θα μπορούσα να αποστείλω πράγματι μια τέτοια συγχαρητήρια επιστολή, γιατί προφανώς ε, ανταποκρίνεται αυτό το ψήφισμα στις επιθυμίες της δικής μας Επιτροπής. Ε, σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ρουμανίας, είπαμε ότι θα συζητήσουμε ε, σήμερα αργότερα για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Γαμά για αυτή την παρέμβαση. Περνάμε τώρα ε, στον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια γνωμοδότηση από την πλευρά τη δικής μας Επιτροπής προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς που είναι της ουσίας Επιτροπή. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου το λόγο γιατί είναι η συντάκτρια της ομοδότησης. Παρακαλώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο αντίκτυπο τη διαφήμιση στη συμπεριφορά των καταναλωτών θα εξεταστεί σε μια ε, έκθεση ε, για ε, την έκθεση του κυρίου Φιλίππου Ιωκυβίνη από την Επιτροπή Ιστορική Αγορά, όπω είπατε, σε ό,τι αφορά την ιστορική αγορά την προστασία των καταναλωτών. Η δική μου λοιπόν συνεισφορά ω συντάκτη αυτή τη γνωμοδότηση για τον αντίκτυπο τη διαφήμιση συμπεριφορά των καταναλωτών από την πλευρά τη Επιτροπή Γυναικών κάνει κάποιες συγκεκριμένες ε, προτάσεις ε, ε, τις οποίες προτείνουμε να περιληφθούν μέσα στην, στο σχέδιο ψηφίσματος. Προφανώς η διαφήμιση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη σημερινή κοινωνία, ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες και προωθεί τον ανταγωνισμό και δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα ανταγωνισμού και δίνει και όθηση στην ε, ενημέρωση με αποτέλεσμα να προωθεί και την ανάπτυξη ε, και να αυξάνει τις επιλογές των καταναλωτών. Ως Επιτροπή FM δεν υποτιμούμε το ρόλο της διαφήμισης σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των ε, απόψεων των συμπεριφορών των καταναλωτών απέναντι σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και λάβουμε, λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη μας τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα φύλλα μέσω των διαφημίσεων. Γι' αυτό ε, πρώτον ε, τονίζουμε ότι η διαφήμιση δεν θα πρέπει να ε, σάγει στερεότυπα σε ό,τι αφορά τα φύλλα, γιατί αυτό βέβαια αποτελεί εμπόδιο στις πολιτικές για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών να έχουν τον νου τους για τέτοιου είδους μηνύματα από την πλευρά των διαφημίσεων. Ταυτόχρονα οι διαφημίσεις δεν θα πρέπει να ε, διαδίδουν κανένας είδου εξιστικά βία ή άλλα μνήματα που προωθούν την ε, άνηση μεταχείριση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την μη αξιοπρεπή ε, προβολή του γυναικείου σώματος. Τρίτον, η διαφήμιση δεν θα πρέπει να προωθεί ένα ιδανικό τελειότητα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το γυναικείο φύλλο αξιοποιώντα έτσι τις ε, αδυναμίες ε, διαφορετικών ομάδων καταναλωτών, ειδικότερα των νέων, και ε, δημιουργώντα προβλήματα όπως η βουλμία η νεορεξία, ειδικότερα σε επαφές ομάδε καταναλωτών. Τέταρτον, η διαφήμιση μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την πρόσληψη τη κοινωνία απέναντι σε ζητήματα όπω ο ρόλο των φίλων, η εικόνα του σώματο και πράγματι μπορεί να συμβάλλει στην θετική απεικόνηση των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία, στον επαγγελματικό του χώρο, στην οικογένεια, στην κοινωνική ζωή. Ε, και πέμπτον, ε, ε, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην έκθεση, εκπαίδευση και στην κατάσταση από την παιδική ηλικία και καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ενδυναμώσουν τις δράσεις εκείνες τις εκπαιδευτικές και κατάρτισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει και μια αυτοδόμηση στον ίδιο τον κλάδο της ε, ε, διαφήμισης ούτως ώστε να υπάρχει μια δεοντολογία στον χώρο της ε, διαφήμισης χωρίς να προωθούνται στερεότυπα και να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των δύο φύλων. Ε, να υπάρχουν διαφημίσεις που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κατά την ε, κατάρτιση της ε, γνωμοδότησής μας είχαμε τον περιορισμό 1500 χαρακτήρων σε ό,τι αφορά δηλαδή το μήκος της γνωμοδότησης, άρα ήμασταν πολύ περιορισμένοι σε ό,τι μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και εγώ θα ήθελα να σας κάνω να υποβάλλετε τις δικές σας ατροπολογίες έως ε, τις 15 Ιουλίου, έως αύριο δηλαδή που είναι και η καταλητική προθεσμία. Η δική μας Επιτροπή θα ψηφίσει επί της δικής ομοδότησης στις 2 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ λέει η πρόεδρος. Και τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιγόνη Παπαδοπούλου γιατί νομίζω ότι στις υποδείξεις της έλαβε υπόψη όλες τις βασικές πτυχές που θα πρέπει να προωθήσει η Επιτροπή των Γυναικών. Σε όλες τις χώρες και ειδικά στην Ιταλία γίνονται πολύ έντονες συζητήσεις για ε, μία εικόνα που προωθείται μέσω διαφημίσεων που ταπεινώνει την ταυτότητα της γυναίκας. Θα προβάλλω και μία πρωτοβουλία στο εγγύς μέλλον, όπου ε, μία σκηνοθέτης Ε, έχει γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πραγματικά είναι μία γροθιά στο στομάχι για το πώς ε, προβάλλεται η γυναίκα και ο ρόλος της γυναίκας. Αυτό θα το προωθήσω στο εγγύς μέλλον. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν και τα ε, κράτη-μέλη να ασχοληθούν εκ νέου με τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό το τομέα με έναν κώδικα συμπεριφοράς και να δούμε πώς αντιμετωπίζουν το όλο θέμα και οι ενώσεις διαφημιστών από πλευράς ε, επαγγελματισμού. Ίσως θα πρέπει να βρούμε ένα πιο αποδοτικό ε, σχήμα, διότι πολλές φορές οι εκκλήσεις μας ε, δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Και θα ήθελα οι γυναίκες να μην αγοράζουν προϊόντα τα οποία διαφημίζονται κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα πρέπει να τα μποϊκοτάρουμε και επίσης να προβάλλουμε οργανούς με ισχυρή παρουσία γυναικών που να έρθουν σε επαφή με χρήστες, με ενώσεις καταναλωτών και να προβάλλουν ένα μηχανισμό εγγυήσεων έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ξανασκεφτούμε και να διορθώσουμε αυτό το πλαίσιο εργασίας. Υπάρχουν συμβουλευτικές επιτροπές, ένας κώδικας δεοντολογίας, ε, οι χρήστες. Ίσως θα πρέπει να προβάλλουμε και εδώ έναν τρόπο διακυβέρνησης, δηλαδή μιλάμε για ε, ελευθερία λόγου, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να προβληθεί ο πραγματικός ρόλος των γυναικών και όχι να προβάλλονται τόσο ταπεινωτικές εικόνες για τις γυναίκες. Και εγώ, θα... θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το γεγονός ότι έχει εστιάσει στα κεφαλαιώδη θέματα που συνάπτονται με αυτό το ζήτημα. Χαίρομαι που η Επιτροπή των Γυναικών έχει προβεί στη γνωμοδότηση αυτή για την, για την επίδραση των ε, διαφημίσεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των γυναικών. Κινδυνεύουμε με τις διαφημίσεις αυτές να διατηρούμε τα στερεότυπα <clears throat> σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και ήταν πολύ θετικό όταν απαγόρευσε η Ισπανική κυβέρνηση μια διαφήμιση της Πράντα διότι είχε παρουσιάσει μια μεγάλη εικόνα μια γυναίκα η οποία είχε γονατίσει σε στάση σκυλιού με έναν άντρα να την κρατάει. Και είπε η Ισπανική κυβέρνηση ότι αυτή η διαφήμιση δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί στην ε, Ισπανία. Η Πράτα, μια Ιταλική εταιρεία, είπε εντάξει αν είναι έτσι εμείς θα αποσύρουμε όλα τα προϊόντα μας από την Ισπανία αλλά και η Γαλλία ακολούθησε το παράδειγμα της ε, Γαλλίας και η Πράντα υποχώρησε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υποστηριχθούν οι προσπάθειες αυτού του είδους και θέλω και εγώ να υποστηρίξω το να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα θέματα αυτά. Και επίσης δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο τα προβλήματα των γυναικών, αλλά γενικά τα θέματα του φύλου. Μπορεί και οι άντρες να παρουσιαστούν με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να είναι επιθετικός και υπήρξε μια δικαστική υπόθεση στη Σουηδία εναντίον μια διαφημιστική εταιρεία που παρουσίασε του άντρε να κάθονται όλη μέρα στου καναπέδε και να μην κάνουν τίποτα. Και αυτό είναι ε, ταπεινωτικό και εναντίον του. <clears throat> Χωρί μικρόφωνο η πρόοδο. Χωρί μικρόφωνο και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως η ε, γνωμοδότηση ε, αποτελεί ε, μία από τις καλύτερες δυνατότητες που έχουμε για να εκφραστούμε, για να διαρευνήσουμε το ζήτημα του τι συμβαίνει στη διαφήμιση και σε σχέση με τις συμπεριφορά σε σχέση με τη διαφήμιση στην Επιτροπή έγινε μια σχετική παρουσίαση χθε σε σχέση με αυτό το ζήτημα και δεν υπήρξε ούτε μία αναφορά στο ζήτημα της ε, μεταχείρισης και της όλης μεταχείρισης μεταξύ των δύο φύλων. Ε, πραγματικά δεν μου άρεσε που δεν υπήρχε καμία αναφορά και γι' αυτό θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να είμαστε ιδιαίτερα κατηγορηματικοί. γιατί τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της διαφήμισης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις ενημερωτικές εκστρατείε, τις οποίες προσπαθούμε να προωθήσουμε, όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει από κοινού με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προκειμένου να αλλάξουμε την συμπεριφορά του ευρέω κοινού. Αυτά δηλαδή που συμβαίνουν στον χώρο της διαφήμισης ουσιαστικά ε, προσπερνούν, δεν λαμβάνουν υπόψη όλα τα, ε, όλες αυτές τις προσπάθειες από τη δική πλευρά και το μόνο που στοχεύουν είναι να προωθήσουν συγκεκριμένα προϊόντα ε, στα και θα ήθελα να πω συγκεκριμένα για τη διαφήμιση όπου έχουμε μία περίπτωση Ε, όπου υπάρχει ένα άντρα ο οποίο καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε μια γυναίκα και σε κάτι άλλο και τελικά επιλέγει το άλλο. Δηλαδή είναι κάτι πραγματικά πολύ ε, μειωτικό για τι γυναίκε και το είδαμε αυτό στο Βέλγιο και νομίζω ότι αλλού υπήρξε αυτή η διαφήμιση και νομίζω πω σωματικά αυτό μα δείχνει ότι θα πρέπει να ε, καταστήσουμε σαφέ ότι τέτοιου είδου τεχνικέ, τέτοιε μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τι δικέ μα πολιτικέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, και σε συνεργασία με την Επιτροπή. Άρα λοιπόν πραγματικά θα πρέπει να είμαστε πολύ κατηγορηματικοί. Ευχαριστούμε πολύ ε, την εισηγήτρια για, για όλα τα σημεία που έλαβα υπόψη στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσα η συζήτηση και στην ουσία πραγματικά της ε, φιλοσοφίας της πολιτικής μας και ήθελα να συγχαρώ και την εισηγήτρια και τη συναδέλφια για τη συμμετοχή τους. Πιστεύω ότι αξίζει να δούμε οι, οι, οι κώδικες δεοντολογίας και οι ασφαλιστικές δικλίδες που υπάρχουν στις διάφορες χώρες, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που αναδύεται το πρόβλημα αυτό, γιατί δεν έχουν αποδώσει και να δούμε τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο της νέας μας ε, προσπάθειας. Διότι δεν είναι πρώτη φορά που αναδύεται το θέμα, ούτε πρώτη φορά που αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το, το Κοινοβούλιο. Και υπάρχουν κώδικες δεοντολογίας, υπάρχουν οργανισμοί που έχουν ευθύνη για την προστασία της αξιοπρέπειας στις χώρες μέλη γιατί δεν έγινε αυτή, αυτό δεν απέδωσε, η αυτορύθμιση που θεωρούσαμε ε, αυτονόητη ε, ότι θα συμβεί δεν έχει λειτουργήσει. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ε, και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και συζήτηση με υπευθύνους από διάφορες χώρες που, έχουν, ε, είναι επικεφαλής αυτών των οργανισμών, κάθε χώρα έχει το δικό της ε, όνομα του αρμόδιου οργανισμού, αλλά πάντα ο στόχος είναι πώς θα σέβονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι διαφημίσεις στην αξιοπρέπεια του ατόμου, γιατί δεν έχουν αποδώσει. Εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί της ε, όλης της ιστορίας, γιατί θεωρητικά κανείς δεν είναι αντίθετος σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Κράτσα. όπως είπε και η κυρία Κράτσα και όπως έχουμε ήδη αναφέρει και στην Επιτροπή μας εγώ έχω παρουσιάσει μια έκθεση πρωτοβουλία σε σχέση με τα θέματα αυτά της επιρροής της ε, διαφήμισης για την συμπεριφορά των καταναλωτών. Και δυστυχώς απεδείχθη ότι και οι γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται από τις διαφημίσεις ότι υπάρχει σημαντική επιρροή των διαφημίσεων στην συμπεριφορά την ανθρώπινη. Η Κομισιόν έχει το λόγο τώρα. Και δεν, είναι παρούσα εκπρόσωπος της Κομισιόν. Δίνω και πάλι το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Νομίζω ότι υπάρχει γενική συνένεση μεταξύ μας ότι η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να δώσει σαφείς κατευθύνσεις προς την αρμόδια επί Επιτροπή. Όλοι έχουν τονίσει ότι τα στερεότυπα των φύλων αναπαράγονται από πάρα πολλέ διαφημίσεις. Και όπως είπε και η κυρία Κώστα, μερικές φορές είναι προκλητικά τα πράγματα ιδίως σε ταινίες και σε μικρά βίντεο, σε κλιπ που παρουσιάζουν τις γυναίκες με ένα τελείως στερεότυπο τρόπο. Οι διαφημίσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κοινωνία των πολιτών και από τις ρυθμιστικές αρχές. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συνεχής διάλογος για τα θέματα αυτά και θα πρέπει να προκύψουν πρότυπα τα οποία θα πρέπει να είναι δεσμευτικά για όλους. Συμφωνώ και με την ιδέα, επίσης, η οποία διατυπώθηκε, ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτές τις στερεότυπες μορφές παρουσίασης των φύλων, ότι αυτό οδηγεί σε διακρίσεις και όπως είπε η κυρία Πανάτοβα, θα πρέπει να δούμε αυτή τη γνωμοδότηση σε μια ευκαιρία να επηρεάσουμε την τελική έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, γιατί σίγουρα <clears throat> θα πρέπει αυτή η έκθεση να τονίσει τον ρόλο των ρυθμιστικών αρχών και των προτύπων που θα προστατεύσουν την εικόνα της γυναίκας. Σύμφωνα και με την κυρία Κράτσα που είπε ότι είναι πολύ σημαντική, σημαντικά τα ηθικά πρότυπα, θα πρέπει να έχουμε τα αποτελεσματικά εργαλεία και τους μηχανισμούς για να εξασφαλίσουμε το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είτε πρόκειται για σώμα ανδρός είτε γυναικός. Γιατί και οι άνδρες την χάνουν διακρίσεων και εκμετάλλευσης επίσης. Και ίσως με τις τροπολογίες μας μπορούμε να πούμε και κάτι για την έρευνα στον τομέα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή μελέτη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες μπορούν να μεταλαμπαδευτούν και ακολουθηθούν από άλλες χώρες. Σε μία από τις προσωπικές μου τροπολογίες λοιπόν θα προτείνω τη δημιουργία τέτοιων μελετών. Δυστυχώς οι γνωμοδοτήσεις περιορίζονται σε 1500 χαρακτήρες. Δεν μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα, είναι τόσα πολλά τα οποία μπορεί να πει κανείς, αλλά στην πράξη μέσα σε 1500 χαρακτήρες μπορεί να πει κανείς ελάχιστα πράγματα και μόνο με τροπολογίες μπορεί να παρουσιάσει την απόψη του. Εγώ θα καταθέσω τροπολογίες και σας λέω και πάλι ότι ακόμα και αν δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι αύριο, ελπίζω ότι όσοι έχουν τροπολογίες θα μας τις δώσουν για να μπορέσουμε να τις προωθήσουμε και αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, <clears throat> κυρία Παπαδοπούλου, για τις προθεσμίες. Αύριο, 15 Ιουλίου, είναι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών μέχρι το μεσημέρι στις 12. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα έρθει το θέμα αυτό και θα ψηφιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου και μάλλον στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου θα περάσει στην ολομέλεια αυτή η έκθεση. Τώρα. Θα ακολουθήσει η ανταλλαγή απόψεων με την αντιπρόεδρο της ε, βελικής κυβέρνησης σε σχέση με τα θέματα αυτά που ασκεί όπως ξέρετε την Προεδρία και περιμένουμε μερικά λεφτά μέχρι να έρθει. Mrs. Pavanova, good. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, meanwhile, while we are... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενώ περιμένουμε, θα ήθελα να προτείνω κάτι διαδικαστικό. Επειδή έχει μεγάλη σημασία η γνωμοδότησή μας ως προς το θέμα της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών, θα ήθελα να πω οι τροπολογίες που θα προβάλλουμε στην έκθεση Παπαδοπούλου να υποβληθούν και στην ΙΜΚΟ για υποστήριξη, διότι πολλές φορές, και λυπάμαι που το λέω αυτό, οι προτάσεις μας αμελούνται. Very Γι' αυτό θα πρέπει να προτείνουμε ε, να υποβάλουμε αυτές τις τροπολογίες και προς τα εκεί. Δεν έχουμε την έκθεση Ζουβά που είναι ο βασικός εισηγητής στην ΙΜΚΟ, αλλά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τακτική για να είμαστε πιο ε, αποτελεσματικοί, αποτελεσματικές. Ευχαριστούμε την κυρία Παρβάνοβα. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ συμμετέχω σε αυτή την επιτροπή και θα είμαι πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες έτσι όπου, εκεί όπου μπορούμε. Αυτό είναι ένας πολύ επικοδομητικός τρόπος εργασίας και σε αυτό το ζήτημα και σε άλλα, έτσι ώστε να αυξήσουμε την επιρροή μας εκεί όπου μπορούμε. Ευχαριστούμε κυρία Πάνοβα για την υπόδειξή σας. På utskottets vägnar så är jag glad att få välkomna från det belgiska Η κυρία Ζωέλ Μιλκέ είναι μαζί μας από την ε, Βελική Προεδρία, είναι αντιπρόεδρος και της Βελικής Κυβέρνησης και υπουργός για την ε, ισότητα των φύλων. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί της σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα της Βελικής Προεδρίας στον τομέα της δικής μας αρμοδιότητος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε σε θέση να πληροφορηθούμε από την κυρία Μιλκέ για τις προθέσεις της Βελγικής Προεδρίας και στη συνέχεια να ανταλλάξουμε απόψεις με, μαζί τη για τα θέματα που μα ενδιαφέρουν. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μιλκέ. Έχετε το λόγο κυρία Υπουργέ. Euh, euh, σα ευχαριστώ πολύ κυρία Σβένσον καθώ και τα μέλη τη Επίτροπή, για την υποδοχή σα ε, και την πρόσκλησή σα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και να σας ε, συναντώ παρακολουθούμε την εξέλιξη της νέας συνθήκης κατά γράμμα και ιδιαίτερα τον νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε αυτή την Επιτροπή, όπως και σε όλες τις άλλες, έτσι ώστε να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε ε, το όλο θέμα από πλευράς της Βελγικής Προεδρίας ή ιδιαίτερα ως προς την ίση πρόσβαση στο χώρο εργασίας ανδρών και γυναικών. Έτσι ώστε να προβάλλουμε και άτυπες συναντήσεις για να τιμήσουμε αυτή την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο γενικότερα. Σε σχέση με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η Βελγική Προεδρία έχει δύο βασικές προτεραιότητες, πολιτικές και νομοθετικές και στο πολιτικό σκέλος προβάλλουμε τρεις άξονες. Καταρχήν να δούμε τις πολιτικές προτεραιότητες και στο τέλος της εισήγησής μου θα απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Για να μιλήσουμε περισσότερο για το νομοθετικό μας έργο μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για την άδεια μητρότητας. Ως προς το πολιτικό σκέλος έχουμε τρεις βασικές προτεραιότητες. Καταρχήν, τον τρόπο ενίσχυσης της πολιτικής απασχόλησης, γιατί ασχολούμε και με θέματα απασχόλησης και νομίζω ότι μπορούμε να προσδώσουμε και αυτή την διάσταση στο θέμα και υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσα στα πλαίσια των στόχων του Πεκίνου. Αυτό ήταν ένα θέμα προτεραιότητας ήδη από το 2001 και θα επανασυνδεθούμε με αυτό το θέμα και θα σας μιλήσω για τις συστάσεις και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στα πλαίσια της χάρτας που προτάθηκε από τη Νέα Επίτροπο εδώ και μερικούς μήνες. Καταρχήν, να υπάρχει ίση πρόσβαση στον, στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος. Είχαμε ε, αγαστή συνεργασία στα πλαίσια της ε, Τρόικας και με τη ε, Βελγική Προεδρία και με τη συνάδελφο Βιβιάνα για να καταπολεμήσουμε και τη βία έναντι των γυναικών. Μετά θα μιλήσω για τα συνοδευτικά μέτρα στα πλαίσια της στρατηγικής ως προς την ισότητα ανδρών και γυναικών που θα προτείνει η Επίτροπος. Καταρχήν, ως προς την ενίσχυση της πολιτικής απασχόλησης και απασχολησιμότητας, ε, εδώ ακριβώς εντάσσεται, και το μισθολογικό χάσμα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή όπου έχουμε τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 με συγκεκριμένους στόχους και μέσα στα πλαίσια μιας συλλογικής δράσης και με άλλους πολιτικούς συνεργούς μπορέσαμε να εντάξουμε στους ε, στόχους και αυτό τον γενικότερο στόχο σε σχέση με το 75% απασχολησιμότητα και τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς την απασχόληση. Μία από τις ε, βασικές ε, προτεραιότητες είναι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 να υπάρξει αύξηση της ποσοστιαίας απασχολησιμότητας. Εάν δούμε τις στατιστικές της Eurostat του Μαρτίου του 2010 βλέπουμε ένα 71% και 58,6% αντιστοίχως για άνδρες και γυναίκες. Και όταν ξέρουμε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής 2020 είναι να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών αυτή θα πρέπει να είναι και η βασική μας ε, στοχοθέτηση για τις γυναίκες και την απασχολησιμότητα των γυναικών. Θα ήθελα λοιπόν αυτή η προτεραιότητα να ενταχθεί στις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης που ενέκρινε το Συμβούλιο της 21ης Οκτωβρίου μέσα στα πλαίσια του εσκό και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε ετήσιες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη πριν από τα προγράμματα αναθεώρησης και θα επανέλθω σημείο προς σημείο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία ως προς τις γυναίκες, όχι μόνο ως προς το δίκτυο απασχόλησης, αλλά και την κατάρτιση καθώς και μέτρα στήριξης και ιδιαίτερα ως προς τη συμφιλίωση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση ως προς τις μελλοντικές πολιτικές μέσα στα πλαίσια και της οικονομικής διακυβέρνησης όπως συγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. σε όλες τις συζητήσεις ε, για θέματα απασχόλησης, είτε πρόκειται για την πράσινη απασχόληση ή την ε, παράταση του προσδόκιμου ζωής θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και αυτή τη συνιστόσα. Δηλαδή μέσα στα πλαίσια της οικονομίας όπου θα γίνεται λιγότερη, μικρότερη χρήση του άνθρακα και στα πλαίσια του κατακαιρματισμού της αγοράς εργασίας θα πρέπει να έχουμε μία στρατηγική ε, συμπερίληψη των γυναικών σε αυτή την στρατηγική διαφορετικά δεν θα συμμετάσχουν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο πολιτικών. Αυτό αφορά και την απασχόληση μέσα στα πλαίσια της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης, διότι οι γυναίκες μεταξύ 55 και 60 ε, έχουν μία απασχολησιμότητα ε, κατά 60%. Της τάξης του 60%. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές ως προς την ποιότητα εργασίας. Και επίσης θα πρέπει να μας απασχολήσει και η επωνομαζόμενη λευκή απασχόληση που αφορά τον τριτογενή τομέα και θα πρέπει να δούμε και την ε, επισφάλεια στην εργασία, στην απασχόληση. Άρα, στις δύο αυτές βασικές συνιστώσεις, ως προς την στρατηγική απασχολησιμότητα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την γύρανση του πληθυσμού και την μετάβαση αυτή, την οικονομική μετάβαση και την, ε, μέσα στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης, όπως ορίστηκε. και στα πλαίσια της Τρόικας και με τη συνάδελφο Βιβιάν είδαμε ότι χρειαζόμαστε μία ε, ποσοστιαία ε, υποστήριξη, δηλαδή αριθμητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τις θέσεις μας, έτσι ώστε και μέσα στα πλαίσια του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ να προωθήσουμε την πολιτική ισότητας ε, της συμμετοχής των φίλων στην αγορά εργασίας. Γιατί η επέκταση της αγοράς εργασίας έχει μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και το πρώτο θέμα σε σχέση με, τις πολιτικές, ε, με την πολιτική απασχόλησης που θα ενταχθεί και στις μελλοντικές μας στρατηγικές. Τώρα, ως προς το μισθολογικό χάσμα που αποτελεί μια προτεραιότητα της Βελικής Προεδρίας με βάση το ψήφισμα της 16ης Ιουνίου του Κοινοβουλίου γιατί προβάλλεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ως προς την ισότητα ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων που ανέρχεται σε 18% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις 24 και 25 Οκτωβρίου θα συνέλθει το Συμβούλιο, το οποίο θα επικεντρώσει την προσοχή του στο μισθολογικό χάσμα, στο μισθολογικό αυτό άνοιγμα, αυτή την ψαλίδα την οποία πρέπει να συρρυκνώσουμε. Και στόχος μας που συμμερίζεται και η Κομισιόν, η οποία θα προβάλλει στον γης μέλλον έναν οδικό χάρτη. Στόχος μας λοιπόν είναι να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να μας δώσουν αριθμητικά στοιχεία ως προς αυτό το μισθολογικό χάσμα έτσι ώστε με ορίζοντα το 2020 να έχουμε ένα άνοιγμα της τάξης του 0 έως 5% το πολύ και όχι 18% όπως έχουμε σήμερα. Και η Συμβουλευτική Επιτροπή Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση αυτού του μισθολογικού χάσματος. Θα συσκεφτούμε με τους κοινωνικούς εταίρους διότι ε, έτσι θα φτάσουμε σε μια διεπαγγελματική συμφωνία στα περισσότερα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε το μισθολογικό. Ξέρετε ότι τα αίτια είναι πολλαπλά για αυτή την μισθολογική ανισότητα για ίση ή παρόμοια εργασία και αφορά στερεότυπα, επαγγελματικά στερεότυπα, κατακαιρματισμό της εργασίας, συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Πρόκειται για οριζόντιες ή ε, εγκάρσιες πολιτικές και θα πρέπει να δούμε πώς ε, όλα αυτά θα τα εντάξουμε σε μία δίκαιη πολιτική αμοιβών, έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι φιλόδοξη ως προς την στρατηγική που θα προβάλλει στο εγγύς μέλλον μέσα στα πλαίσια και της μελλοντικής διάσκεψης για την μελλοντική αντιμετώπιση του μισθολογικού αυτού ανοίγματος. και να προβούμε σε μία συνολική αποτίμηση στα 27 κράτη-μέλη, προβάλλοντας συστάσεις με βάση τους εννέα δείκτες που έχουμε προαποφασίσει και να δούμε κατά πόσο χρειάζονται συμπληρωματικοί δείκτες που θα πρέπει να αναλάβουμε μέσα στα πλαίσια της εποπτείας της πολιτικής απασχόλησης στην ε, εξελικτική πορεία της στρατηγικής 2020. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει και μία διάσταση η οποία λείπει, γιατί λαμβάνουμε υπόψη τις ε, γνωστές αμοιβές, στους γνωστούς τομείς χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη άλλους δείκτες που δεν σχετίζονται με το βασικό μισθό. Δηλαδή υπάρχουν εξομισθολογικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν ε, μια νέα διάσταση για αυτό το άνοιγμα, αυτό το χάσμα. Είναι γεγονός ότι στα πλαίσια αυτής της διάσκεψης θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε φιλόδοξα συμπεράσματα όπως είχε γίνει και στο Συμβούλιο ΕΨΚΟ του Δεκεμβρίου έτσι ώστε να φτάσουμε σε ε, αυτά στοιχεία ε, ως προς συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής διότι οι στόχοι της Βαρκελόνης είχαν ορίσει ένα 90% κάλυψης ε, για τα παιδιά μεταξύ τριών ετών μέχρι το σχολείο και 33% για τις υπόλοιπες κατηγορίες ως προς δίκτυ κάλυψης. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους και μακροχρόνια να τους ξεπεράσουμε εάν θέλουμε να ε, μην φτάσουμε στο 11,5% ε, μείωση συμμετοχής στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες που έχουν παιδιά κάτω από τα τρία έτη. Θα προβάλλουμε λοιπόν συστάσεις και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να ορίσουμε και συγκεκριμένους ε, στόχους, υποκατηγορίες στόχων ως προς την συμφιλίωση ιδιωτικής επαγγελματικής ζωής. Επίσης, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την, ε, τον οριζόντιο αυτό κατακαιρματισμό ή ε, απομόνωση, ιδιαίτερα ως προς τον ε, τριτογενή τομέα όπου οι γυναίκες αμείβονται διαφορετικά. Έχουν χαμηλότερες αμοιβέ. Τρίτος τομέας είναι η... ο κάθετος διαχωρισμός και η ενθάρρυνση των γυναικών να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην επαγγελματική τους ζωή και ιδίως στην επαγγελματική τους καριέρα και στον οικονομικό στίβο. Θέλουμε λοιπόν και στο επίπεδο των ε, θέσεων απασχόλησης που έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, δηλαδή στις κινήσεις προς μία θέση απασχόλησης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την ίδια λογική σε ό,τι αφορά τις κάθετες μετακινήσεις των γυναικών. Ξέρετε ότι οι γυναίκες δεν ξεπερνούν τα 32% σε θέσεις αρχηγών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε δεν ξεπερνούν το 25% σε υψηλές θέσεις δημόσιας θέσης, ούτε το 10% στα διοικητικά συμβουλία των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων, 4% μονάχα των προέδρων των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 0% για τους διοικητές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλος δρόμος να διατρέξουμε. Η Νορβηγία έδωσε ήδη ένα θετικό παράδειγμα γιατί αυτή η χώρα επέβαλε μια ελάχιστη εκπροσώπηση κατά 40% για κάθε φύλλο μέσα στα διοικητικά συμβουλία των επιχειρήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η έκθεσή μα σε σχέση με την ισότητα ανδρών και γυναικών μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης η Επιτροπή <clears throat> για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων έχει υπογραμμίσει το ρόλο της Νορβηγίας και ζήτησε στα κράτη-μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν ε, ε, αποτελεσματικά μέτρα και όχι μονάχα με νομοθετικό τρόπο για να εξισορροπήσουν τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι ένα τομέα που θέλουμε να προωθήσουμε ω Βελική Προεδρία με μεγάλη πεποίθηση, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε μια συνένεση και να μπορούμε να συζητήσουμε καιρό και για δεσμευτικούς στόχους σε ό,τι αφορά την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ είναι ανάγλυφη η θέληση τη Φιλική Προεδρίας για να, να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν για το πρώτο τμήμα των προτεραιοτήτων μα, που είναι η απασχόληση και η διαφορά στι αποδοχές. Μια δεύτερη σημαντική προτεραιότητα που συνδέεται και με την Ισπανική Προεδρία είναι ο αγώνα κατά τη βία που ασκείται κατά των γυναικών. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια σε σχέση με το νομικό πλαίσιο για όλα αυτά, αλλά εμεί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιδιαίτερα σοβαρή προβληματική στις κοινωνίες μας που διατρέχει όλα τα πολιτικά και κοινωνικά ρεύματα και που είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει σε όλες τις χώρες μας. Για να ανταποκριθούμε σε αυτό το στόχο αποφασίσαμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να διοργανώσουμε μια συνδιάσκεψη με την παρουσία και της Κομισιόν που θα οργανώσουμε <clears throat> έτσι από κοινού και θα προσκαλέσουμε και εθνικούς αλλά και ευρωπαίους κοινοβουλευτικούς σε αυτή τη συνδιάσκεψη και ο στόχος μας είναι εκεί να αντιμετωπίσουμε δύο προβλήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Καταρχήν εμείς έχουμε ζητήσει να εκπονηθούν δύο μελέτες για να προετοιμάσουν αυτή τη διάσκεψη που θα χώρα το φθινόπωρο. Καταρχήν να υπάρξει ένας απολογισμός και μία καταγραφή βελτίστων πρακτικών από τις διάφορες εθνικές νομοθεσίε των κρατών μελών μας σε ό,τι αφορά τους κανόνες προστασία και τα μέτρα προστασία και πρόληψης τη βίας κατά των γυναικών. Και εδώ ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα πού βρίσκεται ο υψηλότερο βαθμός προστασίας για τις γυναίκε και να μπορέσουμε επομένως να εξασφαλίσουμε και τη μεταλαμβάνευση βελτίστων πρακτικών και τη συνεργασία στον τομέα αυτό Περιμένουμε πολλά λοιπόν από αυτή τη μελέτη που έχει γίνει από κοινού μαζί με την Κομισιόν. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο μας φαίνεται πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και τις εξελίξεις οι οποίες οφείλονται στην πολιτισμική πολυμορφία των κοινωνιών μας σε όλη αυτή την προβληματική κατά της βίας. Είτε πρόκειται για τους καταναγκαστικούς γάμους και την ε, βία κατά των νεαρών κοριτσιών και όλα αυτά για να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η νομοθετική αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά που αφορούν τη διάκριση κατά των γυναικών και ιδίω τι γυναίκες που προέρχονται από μη ευρωπαϊκές χώρες. για να δώσουμε λοιπόν την κατάλληλη διάσταση σε αυτή την πρωτοβουλία και να δώσουμε συνέχεια στην πρωτοβουλία της Ισπανικής Προεδρίας η οποία ήταν για μας πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήδη είχε παρουσιαστεί αυτό υπό Ελληνική Προεδρία νομίζω το 1992 κάποτε ο στόχος μας ήταν να δώσουμε συνέχεια στην πρωτοβουλία του Κάδηγος που ελήφθη υπό Ισπανική Προεδρία να υπάρξει μια διάσκεψη κορυφής των γυναικών σε θέση ισχύω, ώστε να γίνει αυτή η σύνοδος όλων των γυναικών υπουργών ανεξάρτητα από το χαρτοφυλάκιό τους να έρθουν και να ανταλλάξουν απόψει για τι εμπειρίε τους σε κυβερνήσει κρατών μελών, σε διάφορες θέσει ισχύω και εξουσίας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα τα οποία πολλέ φορέ καλύπτονται από την πολιτική επικουρικότητα. Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση αυτή λοιπόν την προηγούμενη μέρα της μεγάλης συνδιάσκεψης που έχουμε οργανώσει για να αντιμετωπίσουμε και αυτή την προβληματική και για να μπορέσουμε να, ξεπερα... να, δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις στη συνδιάσκεψη αυτή και νομίζω ότι μέσα στη σειρά των επομένων προεδριών θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Είναι χρήσιμο λοιπόν να έχουμε και το συντονισμό και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση μεταξύ των γυναικών στον τομέα της πολιτικής. Τρίτη προτεραιότητα και τελευταία θα είναι το να υποστηρίξουμε την Κομισιόν στην ανάπτυξη της νέας στρατηγικής και του νέου φύλου πορείας για τα επόμενα 4-5 χρόνια για να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την επερχόμενη Ουγγρική Προεδρία υπό την οποία θα εγκριθεί αυτή η νέα στρατηγική πώς θα μπορέσουμε με τα συμπεράσματα της δράσης μας να βοηθήσουμε την Κομισιόν και την Ουγγρική Προεδρία να υποστηρίξει το έργο αυτό. Νομίζω έχουμε ήδη μια σειρά από στόχους στο μυαλό μας που η Κομισιόν θα προωθήσει επί τη βάση της Ευρωπαϊκής Χάρτας που προετοίμασε ήδη η κυρία Ρέντινγκ <clears throat> για όλα αυτά τα θέματα που άπτονται της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, ισότητος αποδοχών, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, αξιοπρέπεια έναντι της βίας που ασκείται σε βάρος τους και επίσης να λάβουμε υπόψη και την εξωτερική διάσταση μας φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να την υπογραμμίσουμε για την ισότητα των φύλων και για την υποστήριξη στις γυναίκες μέσα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς μας στόχους. Τώρα για τις συγκεκριμένες νομοθετικές εργασίες, <clears throat> όπως ξέρετε είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο και ευαίσθητο και έχει να κάνει με την οδηγία για την γονική, για τη μητρική άδεια. Εδώ υπάρχουν κάπως αποκλίνουσες απόψεις ορισμένα σημεία, διαφορετικές τροπολογίες σε σχέση με την πρόταση οδηγίας, την αρχική πρόταση οδηγίας, αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Και εξάλλου αυτή η συζήτηση, η οποία είναι συναρπαστική και εξάλλου θεμητή και απαραίτητη, λαμβάνει χώρα σήμερα σε ένα κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο το οποίο γνωρίζουμε όλοι, το οποίο είναι ιδιαίτερα αρνητικό με πολιτικές λιτότητες στα κράτη-μέλη μας, κάτι το οποίο οδηγεί σε μια διστακτικότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τις πιθανές συνέπειες που θα προκύψουν για τους εθνικούς προϋπολογισμούς με ρυθμίσεις αυτού του είδους. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα ρόλο διευκολυντή ή ενδιαμέσου για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μια κοινή προσέγγιση για τα θέματα αυτά μαζί με το Κοινοβούλιο <clears throat> και στη συνέχεια μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση η οποία θα οδηγήσει στην πρόοδο στα θέματα αυτά υπό Βελγική Προεδρία καλύπτοντας όλες τις απόψεις και να μπορέσουν να συγκεδαστούν οι απόψεις και μεταξύ θεσμικών οργάνων και στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων. Αυτά λοιπόν για τι μεγάλε προτεραιότητε τη Βελική Προεδρίας και είμαι έτοιμη να απαντήσω στη συνέχεια στα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ για τα όσα μας παρουσιάσατε σε ό,τι αφορά τις ε, προτεραιότητες της ε, Βελικής Προεδρίας. Ε, διαπιστώσαμε ότι πράγματι αυτές οι προτεραιότητες στις οποίες θα εστιάσετε ε, ταυτίζονται με τις προτεραιότητες ε, της δικής μας Επιτροπής και έτσι αναμένουμε με χαρά τη συνεργασία μας με τη Βελική Προεδρία. Ο λόγος τώρα εδώ στα μέλη της Επιτροπής μας για να κάνουν τις παρατηρήσεις του κ. Σαραμπέλα πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Εγώ είμαι στην ποσόστοση των ανδρών Είμαστε τέσσερις στους 60 σε αυτή την επιτροπή, αυτή είναι η ανδρική ποσόστοση, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για έναν κοινό αγώνα που ε, προβάλλουμε όλοι μαζί. Χαίρομαι που βρίσκεστε στην ομάδα μας. Εγώ γνωρίζω την ε, ισχυρογνωμοσύνη σας ως προς την στήριξη αυτή της υπόθεσης ισότητα ανδρών και γυναικών. Ε, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία ως προς την επιτυχία του βελγικού προγράμματος. Όμως στην αρχή απογοητεύθηκα στο χώρο που δόθηκε στις γυναίκες ως προς τη διατύπωση των κειμένων, διότι όπως ε, ξέρουμε η Ισπανική Προεδρία έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα προς αυτή την ε, κατεύθυνση και δεν ε, τρέφω πια καμία αμφιβολία αφού σας άκουσα. Θα πρέπει βεβαίως να καταπολεμήσουμε και την βία κατά των γυναικών. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα σε αυτή την Επιτροπή, γιατί και εγώ είχα αναλάβει μία έκθεση η οποία ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου είχαμε 500 ψήφους υπέρ τουλάχιστον και έγινε μια γραπτή δήλωση στη συνέχεια προς τους συναδέλφους των πολιτικών ομάδων. Βλέπουμε λοιπόν ότι την χάνει πλειοψηφία σε αυτή η γραπτή ε, δήλωση, κάτι το οποίο είναι σπάνιο, έτσι ώστε να πιέσουμε και εσείς να επηρεάσετε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργηθεί, ε, να προβληθεί ένα έτος υπέρ των γυναικών και κατά της βίας. Βεβαίως πρόκειται για μια κατάσταση μεταβλητής γεωμετρίας που δεσπόζει στα κράτη. Υπάρχουν αρκετά χάσματα και το ζήτημα ίσως να μην είναι τόσο ευρέως γνωστό μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα. Θα ήθελα να ζητήσετε από την κυρία Ρέντινγκ να αναλάβει αυτό το ζήτημα, να δημιουργηθεί το ένα ε, ε, ευρωπαϊκό έτος για τις γυναίκες τα επόμενα πέντε χρόνια, γιατί το επόμενο έτος είναι αφιερωμένο σε κάτι άλλο. Ένα δεύτερο σημείο εφήγει από εσάς. Χαίρομαι που αναλάβατε την πρωτοβουλία. Ο κύριος Γιάκοψεν, υπουργός ε, της Νορβηγίας, ε, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εγκριθεί αυτός ο νόμος ε, έτσι ώστε ένα 40% των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων απαρτίζεται από γυναίκες. Το 35% δεν είναι αρκετό. Ξεκινάμε όμως από ένα 30% στα εθνικά κοινοβούλια, ανάλογα με τις χώρες, και βλέπουμε ότι αυτό το ποσοστό αυξάνεται μετά από τις εκλογές. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις μιλήσαμε για ένα 10% ως προς τα ανώτερα στελέχη, ως προς τους ε, ε, διοικητές εθνικών τραπεζών έχουμε ένα 0% το 60% των φοιτητών που επιτυγχάνουν στα πανεπιστήμια είναι γυναίκες. Βλέπουμε ε, εδώ δηλαδή ότι υπερεκπροσωπούνται, ενώ στη συνέχεια δεν ισχύει κάτι τέτοιο στο, ε, κατά τη διάρκεια της εργασίας, του εργασιακού βίου. Μιλήσαμε για αναγκαίο κακό, αλλά θα πρέπει να διορθώσουμε αυτή την ποσοστή αναλογία δεσμευτικά τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έτσι ώστε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Δυστυχώς η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα μπορούσαμε να, λάβουμε, να αναλάβουμε θετικές πρωτοβουλίες για να πείσετε του συναδέλφους στα 26 άλλα κράτη-μέλη έτσι ώστε ο νόμος αυτός να είναι δεσμευτικός γιατί αν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις τότε δεν εξελίσσεται και η κοινωνία. Θα ήθελα να μας πείτε τι, ποιες είναι οι προθέσεις σας ως προς, την, προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Μποσκούρτ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Μιλκέ, καταρχήν και να σας θέσω μια σειρά ερωτήσεων σε σχέση με την ε, διάσκεψη που οργανώθηκε από τη Βελγική Προεδρία. Ξέρω ότι είχε διοργανωθεί ήδη στον Οκτώβριο μια συνδιάσκεψη σε σχέση με ορισμένε πρακτικέ όπω ο ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ε, για τα θέματα δικαιοσύνη. Ο στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να καταγράψουμε τις, πα, τις παραδοσιακές αλλά επικίνδυνες αυτές τις πρακτικές και να βρούμε τρόπους να αναχαιτήσουμε αυτές τις πρακτικές. Μου φαίνεται ότι είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προβληματική. Δυστυχώς οι στατιστικές μας δείχνουν ότι το πρόβλημα αυτό οξύνεται στην Ευρώπη και είναι απαραίτητο να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με αποτελεσματικό τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι κατανοώ η διάσκεψη στην οποία αναφερθήκατε έχει <clears throat> αναβληθεί και θα οργανωθεί το Νοέμβριο μια συνδιάσκεψη μόνο για τα θέματα της βίας κατά των γυναικών, επομένως δεν θα συμπεριλάβει αυτές τις παραδοσιακές πρακτικές. Νομίζω ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο μέσα στη συνδιάσκεψη αυτή να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτών των πρακτικών που προανέφερα και αν θα έχουμε επίση τη δυνατότητα να σκεφτούμε για συγκεκριμένε δράσει οι οποίε θα αντιμετωπίσουν αυτέ τι πρακτικέ. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι κατά πόσον αυτή η συνδιάσκεψη που αναφέρεται θα μπορούσε να καλύψει την γενικότερη προβληματική της βίας κατά των γυναικών. Και αν ναι, αν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις ειδικέ αυτές μορφές βίας που οφείλονται σε παραδοσιακές πρακτικές και να δούμε ποια θα ήταν τα μέτρα που δυνητικά θα μπορούσαμε να πάρουμε μαζί με κοινοβουλευτικού και οργανώσει γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Μποσκούρτ. Κυρία Παραβάνοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Υπουργό για την πολύ καλή παρουσίαση που μας έκανε, η οποία ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τα όσα κάνουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή ΦΕΜ. Θα ήθελα να τονίσω δύο ζητήματα εγώ. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη βία, μας είπατε κυρία Υπουργέ πως ε, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, αλλά η δική μας ε, προσέγγιση σε σχέση με αυτή την πρακτική ε, είναι να το αντιμετωπίζουμε ως ένα κοινωνικό θεμελιώδε πρόβλημα και προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε, προσεγγίσουμε ένα τρόπο, αν θέλετε, Διακριτική ε, μεταχείριση. Πάντα προσπαθούμε να το ε, ε, προσεγγίσουμε μέσω της χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι ένα είδο χουλιγανισμού στη Βεβατοκάμαρα. Μιλάμε για την ίση μεταχείριση των γυναικών. Μιλάμε για έναν τρόπο για να βγουν οι γυναίκες από τα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας στην απασχόληση και ούτω καθεξή. Υπάρχουν δηλαδή πολλά είδη βίας ει βάρο των γυναικών πέραν της φυσική βία. Γι' αυτό δεν θα θέλαμε να παραμείνει ο χαρακτηρισμός ε, της βίας μόνο ως η βία σε κερβατοκάμαρο σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, αλλά να ξεφύγουμε από αυτό και να ξεφύγουμε και από τη συζήτηση ε, αν πρόκειται για ζήτημα επικουρικότητα ή όχι, σε ποιανού την αρμοδιότητα ανήκει, να το δούμε ως ένα ζήτημα θεμελιώδους δικαιώματο ε, και ως ένα δικαιώματα, το δικαιώμα των γυναικών το οποίο παραβιάζει στο 15% των γυναικών. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και από την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σε ό,τι αφορά την βία μεταξύ των φίλων και θα θέλαμε να ακούσουμε ποια είναι η δική σας άποψη γιατί δεν έχουμε λάβει ακόμα κάποια σχετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ το Κοινοβούλιο είναι πολύ κατηγορηματικό σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Βλέπω πως ε, έχετε αναλάβει αυτή τη δέσμευση και εσείς προσωπικά και η Προεδρία σας αλλά χρειαζόμαστε την ε, οδηγία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οδηγία, σε ό,τι αφορά την άδεια ε, έχουμε κολλήσει λίγο σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, αλλά το να υπεραπλουστεύουμε το πρόβλημα ως το πρόβλημα κόστους το οποίο προκύπτει κατά την άδεια μητρότητας είναι κάτι το οποίο τελικά υποτιμά τα σχετικά δικαιώματα και το των γυναικών. Ας μην μείνουμε δηλαδή στην επιφάνεια αυτού του, του ζητήματος. Καθώς λοιπόν οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες ε, γεννούν και οι άντρες τουλάχιστον η τεχνολογία το έχει επιτρέψει να κάνουν το ίδιο, θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό το σύστημα περισσότερο από απλά δηλαδή το θέμα του κόστους. Είχαμε μια ε, προκαταρκτική ε, μελέτη και θα ακολουθήσει μία το Σεπτεμβρίο, αλλά η, προκαταρκτική αυτή μελέτη έδειξε ότι δεν υπάρχει πραγματικό, δεν υπάρχει πραγματικό αντίκτυπο στο προπολογισμό. Μιλάμε για ένα αντίκτυπο τη τάξη του 0,000 κάτι στον ε, συνολικό προπολογισμό. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε σε 18 εβδομάδε με βάση το επιχείρημα του κόστου. Ε, το Βέλγιο είναι μία από τι χώρε οι οποίε ε, έχει λάβει εδώ μια ισχυρή στάση. Ε, ξέρω πω απασχολείται η δική σα κυβέρνηση, γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω τη δική σα άποψη σε σχέση με αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας και για τα πολλά ζητήματα που καλύψατε. Ναι, και η δημιουργία θέσεων απασχόληση για τι γυναίκε είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για αυτή την Επιτροπή. Κατά και των περασμένων ετών, εμεί ε, θέσαμε διάφορε εκθέσει ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών ε, ε, εκείνων που έχουν περισσότερο ανάγκη από όλου μια θέση απασχόληση και εκείνε οι γυναίκε είναι εκείνε οι οποίε υφίστανται πολλαπλή και ιδιαίτερα έντονη μεταχείριση. Είτε δηλαδή έχουν βάθρο μετανάστευση, είτε έχουν αναπηρία απειλούνται πολύ περισσότερο με ε, φτώχεια και τα δικά τους ε, προφανώς παιδιά και διάβασα στη δική σας ε, παρουσίαση, δηλαδή την παρουσία της Βελγικής Προεδρίας και το πρόγραμμά σας ότι θα ασχοληθεί και με το ζήτημα της παιδικής ένδυας. Και εκείνο που θα ήθελα εγώ να τονίσω και να θα σας ζητήσω και κατά την δημιουργία του οδικού χάρτη του Roadmap είναι να ε, ε, προωθήσετε και αυτό το ζήτημα. Ούτω ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε σαφείς λύσεις ως προς το πώς θα δώσουμε ε, θέσεις απασχόλησης σε αυτές τις γυναίκες που τις χρειάζονται περισσότερο για τις μητέρες με κατή οικονομική κατάσταση, ειδικότερα στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε πολλέ τέτοιε μητέρε. Ε, μιλάμε για ε, ε μητέρε Ρώμα, ε, οι οποίε το τα παιδιά και οι ίδιε έχουν ξεχωριστή εκπαίδευση. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικών ειδών διακρίσει ει βάρο αυτών των γυναικών. Και σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να φέρουμε και ε, αυτά τα ζητήματα, για παράδειγμα, τον ακροτηρισμό των κοινωνικών ε, γενετικών οργάνων ε, και το ζήτημα της γυναικείας στήρωσης και έχουμε επανειλημμένα καλέσει να εστιάσουμε σε αυτό το ζήτημα καθώς έχουμε δει πολύ καλέ πρακτικές από την πλευρά διαφόρων χωρών οπότε θα θέλαμε πολύ να μας βοηθήσετε να περάσουμε αυτό το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής 2020. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης υπό την Βελγική Προεδρία ως προς το πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτούς τους ε, ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δινή κατάσταση και μένουν σε απομονωμένες ε, ε, διαβιούν απομονωμένα, ούτως ώστε να έχουμε σαφείς κατευθυντές γραμμές μέσα στις, στο 2020. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαρόκα. Η κυρία Κλάς έχει το λόγο. Και μετά την κυρία Κλάς θα δώσω το λόγο στην κυρία Υπουργό για να μπορέσει να απαντήσει στη, στον πρώτο γύρο ερωτήσεων και μετά θα δώσουμε το λόγο σε πέντε ακόμα ομιλήτριες Κράτσα, Τόμσον, ε, Σβένσον και Κώστα. Κύριε Κλάση, έχετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για τις ε, παρατηρήσεις της. Πολλές φορές ε, οι προσπάθειες που γίνονται είναι απλώς σταγόνες εν το ωκεανό. Ελπίζουμε ότι η Βελγική Προεδρία θα μπορέσει να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα αναφερθήκατε στην ε, νέα συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Αποτελεί αυτό λοιπόν πράγματι ένα πραγματικό μοχλό για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ισότητα των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εσείς στη χώρα σας είστε υπεύθυνοι για τα κοινωνικά θέματα και γνωρίζετε πολύ καλά την προβληματική των θεμάτων αυτών που πρέπει να προβληθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε για την ε, παράταση του χρόνου ζωής και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς για κάποιο διαφορετικό πια όριο συνταξιοδότησης, είτε πρόκειται να είναι 68, είτε είναι 70 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι ενδιαφέρουσα και η συζήτηση που αφορά την συνταξιοδότηση των γυναικών σε μια νωρίτερη ηλικία. Είπατε ότι υπάρχει η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα στις αποδοχές. Και εμείς είμαστε φυσικά εναντίον του να υπάρχει διαφορετική ε, πολιτική αποδοχών για ίδια και ίση εργασία. Ποιες είναι οι δυνατότητες όμως που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και πώς συνδέεται αυτό με την παρουσία των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάμε για 40% αλλά πρέπει να μιλάμε για ένα στόχο 50%. Αλλά εγώ αγαπητοί συνάδελφοι είμαι πάντα εναντίον μιας δεσμευτικής ποσόστοσης, μιας υποχρεωτικής τέτοια ρύθμιση. Σκέφτομαι περισσότερο για τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα ανταμείψουν κατά κάποιο τρόπο τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια πολιτική ισότητα στα διοικητικά συμβούλια και στι ανώτερε στελεχικές θέσει. Η προστασία της μητρότητα. Και εδώ θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε. Ποιε είναι οι συγκεκριμένε προτάσεις που θα φέρει η Βελική Πρόεδρε για την προστασία της μητρότητα, εμείς. Περιμένουμε ακόμα την ε, έκθεση αντικτύπου και εγώ δεν συμφωνώ με την κυρία Παρβάνοβα που, έχω, που είπε ότι έχουμε ήδη τα στοιχεία Έχουμε κάποια στοιχεία, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε η σωστή προσέγγιση. Όπως ξέρετε, έρχομαι από τη Γερμανία και η Γερμανία πάντα δίνει μεγάλη σημασία να καταγραφεί και να εξεταστεί η τωρινή κατάσταση των καθεστώτων προστασία στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με την προστασία, παραδείγματος χάρη, των, ε, των ε, μάλλον τη δυνατότητα αγωνικής άδεια και τη δυνατότητα προστασίας της μητρότητας της χώρα μας. Κατά τη δική μου άποψη λοιπόν, και πιστεύω ότι το συμμερίζονται αυτό πολλοί συνάδελφοι εδώ στην ε, Επιτροπή μας, θα πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος ε, γαλουχίας κατά κάποιο τρόπο των παιδιών, ένας χρόνος ο, ο οποίος θα πρέπει να είναι προς το πλήρες όφελος της μητέρας και να μην οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα μετά στον χώρο εργασίας. Γιατί πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο οι γυναίκες να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους όταν λαμβάνουν μια σημαντική μητρική άδεια. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι αυτά τα οποία θα προτείνει η Βελική Προεδρία για την προστασία της μητρότητος θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια σωστή και ισορροπημένη έκθεση αντικτύπου για τα θέματα αυτά και ελπίζουμε ότι θα πάρετε τις απαραίτητες επαφές με τα κράτη-μέλη για να μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση και να έχουμε μια καταγραφή των καταστάσεων σε αυτά τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κλάς. Ξαναδίνω το λόγο στην κυρία... Θα δώσω το λόγο μάλλον στην κυρία Κράτσα πριν απαντήσει η κυρία Υπουργό. Κυρία Κάτσα, έχετε το λόγο. Και θα είμαι σύντομη. Κυρία Υπουργέ, ε, παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλε τι διαστάσει του προγράμματο που μα ξεδιπλώσατε και εύχομαι καλή επιτυχία στο στόχο σα. Ακόμη μια φορά ενώνουμε τη φωνή μα με την Προεδρία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ακριβώς γιατί θέλουμε να, πετύχουν, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των στόχων. Εγώ θα σταθώ στο θέμα της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Είναι μια καλή συγκυρία αυτό για την Επιτροπή μας, διότι ήδη έχει εγκριθεί μια έκθεση πρωτοβουλία σε ένα αίτημα που υπέβαλα προσωπικά και θα έχω την τιμή να παρουσιάσω μια πρόταση ψηφίσματος και γι' αυτό το λόγο διοργανώνουμε και μια δημόσια ακρόαση ε, το Σεπτέμβριο για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας επισήσω την προσοχή ότι θα πρέπει να δούμε περισσότερο τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε κι εσείς, αναφερόμαστε συνήθως και ο τύπος και εμείς στο ε, νορβηγικό μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά έχει, αρχίσει, έχει λειτουργεί ήδη. Αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και νομοθετική πρωτοβουλία στη Γαλλία και πολιτικός διάλογος και κοινοβουλευτικός διάλογος για το θέμα αυτό και αρχίζει μια συζήτηση από τα κρατήδια της Γερμανίας για να φτάσει στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, εμείς η δημόσια κρόαση, στην πρόταση που θα υποβάλει η πολιτική μου ομάδα, είναι να εξετάσουμε αυτές τις ε, ε, πρωτοβουλίες που ε, σήμερα είναι υπό επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προσκαλέσουμε και εσάς αυτή τη δημόσια κρόαση να μας πείτε σε ποιο επίπεδο ρήμανσης είναι η πρωτοβουλία της Βελγικής Προεδρίας και ευχαριστώ που το έχετε στις προτεραιότητές σας. Απλά δεν υποβάλλω ένα αίτημα, απλά υπενθύμηση ότι υπάρχει συζήτηση πολιτική και κοινοβουλευτική στην Ευρώπη και πρέπει να την αξιοποιήσετε και εσείς και εμείς σε αυτή τη συγκυρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Κράτσα. Δίνω το λόγο στην κυρία Υπουργό. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε στα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Έχετε το λόγο λοιπόν για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που υποβλήθηκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στους πάντες ε, εντάχει, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα για τα καλά σας λόγια και εγώ είμαι υπέρμαχος της ιδέας ε, της αφιέρωσης ενός έτους στην καταπολέμηση της βίας, ιδιαίτερα κατά των γυναικών. Έχουμε προγραμματίσει με την κυρία ε, Ρέντινγκ μία συνάντηση πριν από την εκπόνηση αυτής της στρατηγικής, της γενικότερης στρατηγικής. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι μία ημέρα μέσα στο έτος ή ένα έτος ολόκληρο αφιερωμένο στην καταπολέμηση της βίας ως προς τις ποσοστώσεις, αυτή τη συλλογιστική, όπως είπε και η κυρία Κράτσα, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να θίξουμε αυτό το θέμα, διότι υπάρχει μεγαλύτερη ενσυνειδητότητα ως προς το θέμα και μέσα στα πλαίσια της οικονομικής ε, διακυβέρνησης επίσης έχουν εκπονηθεί μελέτες για την οικονομική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και ε, το όλο ζήτημα συνδέεται στο ότι συμμετέχουν γυναίκες στο διοικητικό, στα διοικητικά συμβούλια ή είναι ανώτερα στελέχη. Υπάρχει δηλαδή σύμφωνα με μελέτες αυτή η αιτιώδη συνάφεια και είναι κάτι το οποίο θα προωθήσουμε στο μέλλον και στον τομέα της πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης. Θα έρθουμε σε επαφή με την Επίτροπο για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα στα πλαίσια της μελλοντικής στρατηγικής και πρόθεσή μου στα πλαίσια της Προεδρίας είναι να συγκεράσω αυτές τις απόψεις και να δω κατά πόσο στο μέλλον μπορούμε να επιτύχουμε μία συνένεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση τις δικές σας υποδείξεις και υποστήριξη για να είμαστε σαφείς στα συμπεράσματα στα οποία θα φτάσουμε το Δεκέμβριο και να έχουμε μία συνενετική εκούσια προσέγγιση ως προς αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ως προς την οικονομική διακυβέρνηση, αυτή η συζήτηση γίνεται όλο ένα και πιο ανοιχτή, ιδιαίτερα σε τομείς που δεν δεσπόζει η γυναικεία παρουσία. Θα δείξουμε αυτό το θέμα σε εκούσια βάση, σε θελούσια βάση, μέσα στα πλαίσια των ε, συμπερασμάτων στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Ως προς αυτά που ανέφερε η κυρία Μπόσκουρτ, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ε, στα πλαίσια της διάσκεψης. Ε, προετοιμάσαμε αυτή την Προεδρία με την Κομισιόν λάβαμε υπόψη ορισμένες ημερομηνίες ορόσημα. Αλλά αντί να γίνει 8 Οκτωβρίου θα γίνει 25-26 Νοεμβρίου αυτή η, η διάσκεψη. Στις 24 θα συναντηθούν οι γυναίκες υπουργοί και ελπίζουμε να έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε και με τις ανταλλαγές χρηστών πρακτικών και να δούμε και την αυτή θεματική ως προς τις παραδοσιακές ε, πρακτικές, ε, νέες μορφές βίας, ε, διαπολιτισμικά στοιχεία, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα εγκλήματα τιμής, οι ακροτηριασμοί και ούτω καθεξής. Πρόκειται για θέματα που δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς. Άρα στη διημερίδα αυτή θα ακούσουμε και εμπειρογνώμονες. Έχουμε και δύο μελέτες ως προς αυτή τη νέα συλλογιστική και πώς αντιδρούν τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια συστάσεων. Δεν αρκούν τα παχιά λόγια. Θα πρέπει στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου να έχουμε και συγκεκριμένες συστάσεις ή να δώσουμε μία συνέχεια σε αυτές τις διαδικασίες. Για την κυρία Παρβάνοβα θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι τις ιδέες της και εγώ είμαι νομικός και ξέρω ότι γίνεται μια συζήτηση ως προς τη νομική βάση που σχετίζεται σε θέματα ε, διαχωρισμού των φύλων, θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε μία οδηγία για να δούμε το θέμα της βίας και να κινηθούμε προς μία εναρμόνιση. Να είμαστε σαφείς ως προς την ε, νομική ε, βάση. Εν πάση περιπτώσει, συμμερίζομαι αυτές τις ιδέες. Αναφερθήκαμε και στο θέμα της άδειας μητρότητος και εδώ μπορώ να απαντήσω στην κυρία Κλάς. Προφανώς δεν πρέπει να περιορίσουμε όλη την προβληματική ναι. της, ε, της άδειας μητρότητος σε χρονικά και μόνο όρια. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ε, καταβολή των αντιστοίχων από επιδομάτων στις, ε, στις γυναίκες οι οποίες είναι επίτοκες δεν πρέπει να περιορίσουμε όμως το θέμα αυτό μονάχα στα πλαίσια της, της συζήτησης για τα οικονομικά θέματα. <clears throat> τα αναφέρω αυτά ως, ε, ε προ, ως ε, της Προεδρίας, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες στα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά. Εγώ δεν θέλω να μπω μονάχα σε μία αντιμετώπιση που λέει ότι εφόσον υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο προπολογισμού θα τα βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα στο ψυγείο. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μία ενδεχόμενη συνένεση ή να φτάσουμε σε νέες προτάσεις. Υπάρχουν πολλές προτάσεις και τροπολογίες και του Κοινοβουλίου που ε, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς να μην υποσκάψουμε όμως, να μην υποβαθμίσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες στα πλαίσια των μελλοντικών συζητήσεων. Τι θα πρέπει να επιλέξουμε ως στοιχεία για μια μελλοντική στρατηγική και να δούμε και τις τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης και Επιτροπής Γενεκών για να κρατήσουμε την ουσία και να προβάλλουμε ε, σε 20 εβδομάδες κάτι το συγκεκριμένο. Μια πρόταση από την Επιτροπή και την Επιτροπή Απασχόλησης. Εγώ θέλω να προωθήσουμε τα πράγματα και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μην οροδούμε και να προωθήσουμε έναν τριμερή διάλογο για μια απότερη συνένεση. Ε, Madame Ως προς την κυρία Ζαλόφκα, δεν θα πρέπει, θα πρέπει μάλλον να προωθήσουμε το θέμα της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, δηλαδή να προβούμε σε διασταυρώμενους ελέγχους για να εντοπίσουμε αυτές τις διακρίσεις και να δούμε αυτές τις διασταυρούμενες διακρίσεις εκεί που υπάρχουν έτσι ώστε να προωθήσουμε και ε, μία οδηγία για την καταπολέμηση των ε, διακρίσεων και εκεί υπάρχει το θέμα των διασταυρούμενων διακρίσεων. Ε, δυστυχώς έχει μείνει πίσω αυτή η οδηγία. Καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φτώχειας με τον ε, συνάδελφο που ασχολείται με θέματα καθαρά κοινωνικά και απασχόλησης. Προς την κυρία Κλάς πώς ε, μπορούμε να ε, καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα μισθολογικά χάσματα, πώς μπορούμε να προβάλλουμε μία μόχλευση ως προς τα οχάσμα αυτό το μισθολογικό. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να αναλάβουμε δεσμεύσεις και σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε επίπεδο Βελγίου, γιατί εάν δεν ε, επιτύχουμε διεπαγγελματικές συμφωνίες ή τουλάχιστον ατομεακές, δεν θα μπορέσουμε να ενταχθούμε σε αυτή την λογική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Σε σχέση τώρα με την κυρία Κράτσα, νομίζω ότι σας απάντησα. Γνωρίζω ε, πόση και ποια εργασία έχει επιτελεσθεί. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις άλλες ερωτήσεις. Ε, δεν έχουν παραμείνει κενά ή αναπάντητα ερωτήματα. Καλώ συνεχίζουμε λοιπόν με τον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Χιμένε έχει. <laughs> Muchísimas gracias. He escuchado con muchísima. Άκουσα με, μεγάλη, με μεγάλο ενδιαφέρον τις ε, προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας και θα ήθελα να σας συγχαρώ διότι θίξατε ένα θέμα ύψης της ε, σημασίας για τις γυναίκες. Εγώ προέρχομαι από την Ανδαλουσία όπου υπάρχει ένας υψηλός δείκτης ανεργίας και η ανεργία στις γυναίκες είναι πολύ υψηλή, φτάνει ένα 30%. Πολλές φορές ακούω ερωτήματα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Δηλαδή να δούμε την ανεργία των γυναικών και να την αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα. Δεν θα επιμείνω. Αφορά τη βία στα πλαίσια των δύο φίλων, επειδή είμαι η για μια κοινή έκθεση με την κυρία Κάρμεν Ρομέρο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα εντολή, Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η απόψή σας. Θα έρθουμε σε επαφή και με εκπροσώπους της Βελγικής Προεδρίας για να δούμε κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εργασία. Η Ευρωεντολή αντιμετώπισε θέματα, ε, προσέκρουσε μάλλον σε θέματα αρμοδιοτήτων για το πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε τις νομοθεσίες ως προς το αστικό και το ποινικό δίκαιο. Όμως είναι κοινό στόχος και θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτόν, διότι το θέμα της βίας από τα δύο φύλλα είναι ένα θέμα που θα πρέπει να τύχει ευρωπαϊκής αντιμετώπισης από πλευράς Ισπανίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τάχιστα το θέμα, θα πρέπει να έχουμε κοινή αντιμετώπιση γιατί το θέμα γίνεται όλο ένα και πιο περίπλοκο. Σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας για τις 26 Νοεμβρίου, για αυτή τη διάσκεψη. Θα ήθελα να συνεργαστώ και εγώ μαζί σας, γιατί μίλησα, μίλησαμε και με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα ε, γενετικών ακροτηριασμών, εγκλημάτων τιμής και ε, ε, γάμων και llegan a καταναγκαστικούς ε, γάμους και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, μην οροδίσουμε διότι υπάρχουν θέματα καθαρά θρησκευτικά και θέματα ε, αστικού και ποινικού δικαίου τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ως προς το θέμα της, της ένδυσης θα πρέπει να δούμε τι στάση θα... Σας ευχαριστώ. Κύριε σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εντυπωσιάστηκα πολύ από το φιλόδοξο πρόγραμμά σας ε, για την ισότητα, γιατί δείχνει να καλύπτει όλους ε, ε, τους τομείς στους οποίους εργαζόμαστε στη δική μας Επιτροπή και τομείς οι οποίοι έχουν σκοπό να βελτιώσουν την ισότητα μεταξύ των ε, δύο φύλων στην Ευρώπη. Και επίσης η δική σας προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας είναι πολύ ε, μοντέρνα, πολύ σύγχρονη, γιατί σημαίνει ότι θα έχουν περισσότερες ευκαιρίε, ε, θα έχουν πιο ισότιμη μεταχείριση έχοντα πλήρη πρόσβαση στην ε, αγορά εργασία οι γυναίκε και από την άλλη πλευρά όπως μας είπατε, το χαρακτηριστικό μιας υγιούς κοινωνίας είναι το να εργάζονται όσο γίνεται περισσότερα μέλη της. Ε, επίσης μου άρεσαν ε, τα ε, όσα, ε, όσα είπατε σε σχέση με τα διοικητικά συμβούλια και τη συμμετοχή των γυναικών και της, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την έννοια των πρασίνων θέσεων εργασίας και το πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε περισσότερες δεξιότητες ε, ε, για γυναίκες ούτως ώστε να ε, απασχολούνται και σε αυτόν τον τομέα των φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών. Όλα λοιπόν αυτά μου φαίνονται πολύ προοδευτικά. Αλλά σε ό,τι αφορά την μισθολογική διαφορά ανδρών και γυναικών, ε, μας είπατε και σωστά έχετε τους λόγους σας, κάτι που εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να δούμε την ε, οδηγία για την άδεια ε, σε σχέση με αυτό το ζήτημα της μισολογικής διαφοράς. Δηλαδή, εμείς θέλουμε περισσότερα παιδιά στην Ευρώπη λόγω του δημογραφικού μας προβλήματος. Κατά συνέπεια, θέλουμε να έχουμε περισσότερα παιδιά. Αλλά αυτό που βλέπουμε από όλες τις στατιστικές της ε, Eurostat είναι ότι αυτή η μισολογική διαφορά ε, παρουσιάζεται όταν οι γυναίκες γίνονται μητέρες. Εκεί μειώνονται οι μισθοί και εκεί αυξάνεται η διαφορά. Ενώ μειώνεται η διαφορά όταν είναι στην ίδια κατάσταση οι γυναίκες με τους άντρες. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αν δεν υπάρξει σωστή κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων μέσα στην οικογένεια, δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ το πρόβλημα τη μισολογική διαφορά. Δηλαδή ένα βασικό πρόβλημα εδώ είναι ότι οι γυναίκε είναι αρμόδιες για τα παιδιά. Και είναι σημαντικό από σε 17 κράτη-μέλη έχουμε και την δυνατότητα άδεια πατρότητα ε, για του πατέρε ε, δηλαδή. Ε, όχι βέβαια τη ίδια διάρκεια, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ω θεσμό. Και προφανώς αυτή η αντιμετώπιση θα πρέπει να ισχύει τόσο για του άνδρε όσο και για τι γυναίκε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αυτή η διακριτική μεταχείριση ό,τι αφορά του γονεί θα συνεχίσει να υφίσταται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η άδεια που θα περιλαμβάνει και τουλάχιστον τη εβδομάδα στα πατρότητα για τον πατέρα ή να υπάρξει ακουστή οδηγία για την άδεια πατρότητα, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και σχετική πρόθυμη από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν πάντα ε, πηγαίνουμε στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή ε, σε επίπεδο Ευρώπης, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί δηλαδή πάντα να, ό,τι αποφασίζουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο, κάτω από το στάδιο το οποίο τηρούν τα κράτη. Θα ήθελα λοιπόν να κάνετε και τη σχολεία σε ό,τι αφορά την αδιαμετρότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμσον. Και εγώ ζήτησα το λόγο για να μιλήσω για το θέμα αυτό και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Κώστα. Εγώ εξετίμησε ιδιαίτερα τις προτεραιότητες που διαγράψατε στα θέματα της απασχόλησης ως Βελγική Προεδρία. Νομίζω ότι τονίσατε τη σημασία της ε, απασχόλησης των γυναικών για να εξασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών. Θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η καλύτερη πλατφόρμα για την ισότητα ευκαιριών, δηλαδή οι γυναίκες να έχουν την πρόσβαση στην αγορά εργασία και να έχουν τη δυνατότητα να είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν για τις γυναίκες να έχουν μια πραγματική ισότητα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βρουν εργασία οι γυναίκες. Να υπάρχουν συστήματα τα οποία επιτρέπουν την φροντίδα των παιδιών και επίσης των ηλικιωμένων η επίτευξη των στόχων της Βαρκελόνης όπως είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν και διαπιστώνουμε ότι η στόχη αυτή της Βαρκελόνης δεν επιτέθησε. Και γι' αυτό θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι νέες πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν από τη Βελική Προεδρία για να γίνουν σεβαστοί οι στόχοι αυτοί σε ό,τι αφορά την παιδική φροντίδα, τους βρεφονιπιακούς αθμούς, και για το θέμα της μητρικής άδεια. Εγώ μιλώ περισσότερο για γονική άδεια, γιατί και οι δύο ομού γονείς θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ανατροφής των παιδιών. Και η μητέρα και ο πατέρας. Και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της Βελικής Προεδρίας θα <clears throat> υπάρξει και μια απόφαση σε ό,τι αφορά την μητρική μάλλον γονική άδεια Και επομένω θα ήθελα να ξέρω ποιε είναι οι πρωτοβουλίε σα στον τομέα αυτό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τη δυνατότητα αύξηση τη απασχόληση των γυναικών και να κατανοήσουμε και ποια είναι τα ωφέλη τα οποία θα προκύψουν από μια ευρύτερη απασχόληση των γυναικών. Και χρειάζεται επίσης να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπου το επίπεδο συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών και των ανδρών βρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο. Και εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν οι ρυθμίσεις για την φροντίδα των παιδιών και για τη γονική άδεια. Ενώ τούμπαλιν στις χώρες όπου η απασχόληση των γυναικών είναι είναι υποδέστεροι εκεί που ελείπουν αυτά τα κοινωνικά συστήματα η μέρημνα των παιδιών και των ηλικιωμένων και η γονική άδεια. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Κώστα και μετά στην κυρία Υπουργό για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερα την παρέμβαση της Υπουργού και θα την ήθελα να την ευχαριστήσω για την σαφήνειά της ως προς την προβολή ορισμένων συγκεκριμένων στρατηγικών της βελικής αντιπροσωπείας. Και θα ήθελα να λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μία συγκυρία όπου επιδεινώνεται η χρηματοπιστωτική κρίση, αυξάνεται η ανεργία και γίνονται περικοπές από τα κράτη-μέλη, τα οποία κράτη-μέλη περικόπτουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτά τα θέματα και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε μια διπλή πρόκληση την πρόκληση της κρίσης, γι' αυτό θα πρέπει να εποπτεύσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις της ε, κρίσης κατά των γυναικών και παράλληλα την προοπτική της Ευρώπης 2020, όπου η προσέγγιση των φύλων, της ισότητας των φύλων δεν έχει βαθυνθεί επαρκώς. Άρα θα πρέπει να μιλήσουμε για συγκεκριμένες δράσεις, αλλά να δούμε και το mainstreaming, την ίση προσέγγιση, έτσι ώστε να προβάλλουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο όπου οι γυναίκες να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο. Δέχομαι την προσέγγισή σας ως προς αυτό το μισθολογικό χάσμα. Νομίζω ότι το μισθολογικό χάσμα ε, θα πρέπει να ε, λαμβάνει υπόψη ότι ο βασικός μισθός είναι ο ίδιος, διότι αυτό αφορά τις συλλογικέ συμβάσεις, ενώ ε, διευρύνεται η ψαλίδα ως προς άλλες εργασιακές βάσεις ή συμβατικές βάσεις. Γι' αυτό αυτή η πρωτοβουλία του Οκτωβρίου θα πρέπει, σε αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει να ε, προηγηθεί ένα ερωτηματολόγιο προς τα κράτη-μέλη ως προς αυτό το σκέλος, διότι δεν έχουμε όλες τις παραμέτρους για να ξέρουμε πού είναι τα προσκόμματα επακριβώς. Γι' αυτό ε, συμμερίζομαι την ε, πραγματιστική σας προσέγγιση. Ως προς τις νέες μορφές ε, βίας, δεν φορούν μόνο τους μετανάστες. Υπάρχουν μορφές βίας που σχετίζονται και από το, τον ας το πούμε εκπολιτισμένο κόσμο. Δηλαδή ε, υπάρχει βία που προβάλλεται και από τα ΜΜΕ, ψυχολογική βία, η οποία πλήττει τη γυναικεία ταυτότητα. Το stalking, για παράδειγμα, έχει μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να δείτε, να λάβετε υπόψη ότι η Ιταλία προέβαλε πρόσφατα μία νομοθεσία και ε, σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζεται και αυτή η νέα μορφή δουλείας που προωθεί το ευρωπαϊκό έγκλημα, τα ευρωπαϊκά δίκτυα εγκλήματος. Και ελπίζω η Βελγική Προεδρία να λάβει υπόψη αυτή την ε, ε, γνωμοδότηση ε, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη αυτή την υποστηρικτική βάση και ως προς ένα τελευταίο σημείο. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι η χορήγηση ε, ηθαγένειας στους ε, μετανάστες. Όπως είπατε, πολύ σωστά στο έγγραφό σας υπάρχουν ε, διαφορετικές προσεγγίσεις από τα κράτη-μέλη. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπου χορηγείται υπηκότητα τα παιδιά που γεννιούνται σε Ιταλικό έδαφος και λαμβάνουν την υπηκότητα όταν συμπληρώσουν το 18ο, το 18 με συγχωρείτε, έτος της ηλικίας τους, ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πώς βλέπετε αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ κυρία Κώστα και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Υπουργό για να δώσει πλήρες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα τα οποία Σας ευχαριστώ πολύ. απαντών καταρχήν στην κυρία Χιμένες και εμείς φυσικά συμμετέσχαμε σε αυτή την πρόταση που αναφέρατε, στην πρόταση οδηγίας και η οποία είναι θετική και υποστηρικτική του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για την Προστασία των Θυμάτων. Νομίζω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας μου έχει παρουσιάσει το θέμα αυτό στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν ίσως κάποιες δυσκολίες, αρμοδιότητες σε επίπεδο ευρωπαϊκό, όπως και σε πολλές χώρες. Η διάσταση του φύλου και η νομική διάσταση πολλές φορές επικαλύπτονται. Αλλά εμείς ως Βελική Προεδρία έχουμε την πρόθεση να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Ακολουθώντας και το παράδειγμα της Ισπανικής Προεδρίας. Και αυτός είναι και ο στόχος της συνδιάσκεψης που θα οργανώσουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε στο φως αυτήν την προβληματική. Μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικής ε, προβληματικής που έχει να κάνει με την βία. Είμαι στη διάθεσή σας λοιπόν για να συζητήσουμε περαιτέρω, να οργανώσουμε αυτά τα θέματα και όπως είπατε επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε το σύνολο της ειδικότερης προβληματικής που έχει να κάνει με τις ε, με τις νέες γυναίκες που, ή τις λιγότερο νέες γυναίκες που έχουν προέλευση από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την κυρία Τόμσεν και εγώ υποστηρίζω να μιλάμε και για πατρική άδεια. Και χαίρομαι για την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έλαβε υπόψη αυτή την πτυχή, γιατί έτσι ξεκινάει μια πραγματική ισότητα να μοιράζονται οι γονείς και την ευθύνη της φροντίδας και της παιδείας των παιδιών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προωθήσουμε στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Για την κυρία Σβένσον, η οποία είπε κάτι σχετικό με όλα αυτά, Θα μπορούσε λοιπόν η έννοια της γονικής άδειας να είναι ευρύτερη από την μητρική άδεια και θα μας, επιτρέ... επέτρεπε να έχουμε αυτή την ευρύτερη αντιμετώπιση και εξάλλου υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν πρόσφατα αναλυφθεί και τις οποίες θα πρέπει να τις προωθήσουμε έτσι περισσότερο βολονταριστικά και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε για τους στόχους της Βαρκελόνης και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την υποδοχή και την φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων και που συνδέονται με την παρουσία των γυναικών στον χώρο της εργασίας. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη με πιο μεγάλο ειδικό βάρος αυτό το θέμα σε όλα τα επίπεδα απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του θέματος είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το Συμβούλιο για τα κοινωνικά θέματα, με όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε και τους επιμέρους στόχους με στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε πιο δεσμευτικές συστάσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών και μετά από αυτή τη συζήτηση τελικά αυτό είναι το πιο σημαντικό να αντιμετωπίσουμε και την ε, προβληματική της νέας οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε πριν από τα γενικά συμπεράσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πριν από τις συστάσεις που εγκρίνονται σε εθνική βάση μετά από την κατάθεση των εθνικών προγραμμάτων, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σαφείς συστάσεις και πιο στοχευμένους στόχους. Αυτά όλα οδηγούν σε μια δυναμική η οποία θα αντιμετωπίσει καλύτερα τους στόχους ισότητας των γυναικών και της βελτίωσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο σε συνεργασία και για την κυρία Κώστα μιλήσατε για την ενσωμάτωση διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο mainstreaming, και θα μιλήσω με την κυρία Ρέντινγκ για το θέμα αυτό. Με την Ουγγαρία το Βέλγιο ζήτησε να δοθεί μια πιο εγκάρσια διάσταση σε όλα τα θέματα που άπτονται του φύλου και να λάβουμε υπόψη παραγωγικά τη σύνδεση με θέματα ανταγωνιστικότητος. Ζητήσαμε στα θεματικά συμβούλια τα οποία προτείνονται από τη Νέα Προεδρία, όπω παραδείγματο χάρη για την έρευνα, ίσω όχι υπό την τρέχουσα Προεδρία, αλλά για την επερχόμενη Προεδρία, να προσπαθήσουμε να δούμε πώ μπορούμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό θεματικό συμβούλιο για τη διάσταση του φύλου και τη σύνδεση με την ε, ε, οικονομική διακυβέρνηση και την Ευρώπη του 2020. Εγώ, επομένως, συμμερίζομαι το όραμά σας, το οποίο είναι ευρύτερο και δεν περιορίζεται μονάχα στην εξασφάλιση ίσων αποδοχών. και υποστηρίζω πλήρως και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη συνδιάσκεψη των δύο ημερών για τη βία. Όχι μονάχα η σωματική βία. Όχι, φυσικά είναι σημαντική η σωματική βία. Αλλά και την βία που ασκείται μέσα στις χώρες μας. Βλέποντας αυτά που γίνονται στις χώρες μας είναι δύσκολο να δώσουμε διδάγματα σε άλλες χώρες. Αλλά να περάσουμε από την σωματική απλώς βία και να περάσουμε στην πιο ευρύτερη μορφή βίας που είναι η παρενόχληση, η ψυχολογική βία, η λαθρεμπορία ανθρωπινών όντων, και αυτό θα το αντιμετωπίσει η Βελική Προεδρία και όλα αυτά συνδέονται. Για την τρίτη σας παρατήρηση, επίσης είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη και τα θέματα που συνδέονται με τη μετανάστευση, πέρα από το ζήτημα της ε, απασχόλησης, με ενδιαφέρει το να επιτύχουμε μια πραγματική πολυπολιτισμική κοινωνία. Και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε να έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες θα καλύψουν και αυτή τη διάσταση, ακολουθώντας και αυτά τα οποία έκανε στην Σαραγώσα η Ισπανική κυβέρνηση. Προεδρία. Υπάρχουν επίσης οι αναλύσεις του ΟΣΑ σε σχέση με τον αντίκτυπο της ε, απόκτησης ηθαγένειας ατόμων από τρίτες χώρες για την αγορά εργασίας και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό το θέσαμε σαν μια από τις κύριες προτεραιότητές μας στην διάσκεψη για την ισότητα όπου θα μιλήσουμε και για την πρόσβαση στην αγορά εργασία ατόμων από τρίτε χώρε και φυσικά είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο των γυναικών εκεί πέρα. Αυτά. Θα ήθελα να σα πω, κυρία Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ. Jag vill framföra utskottets varma tack. Ε, εξ ονόματος της Επιτροπής μας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την επίσκεψή σας σήμερα στην Επιτροπή μας και για το ενδιαφέρον που δείχνει η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου και προφανώς αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνεργασία μας με την Προεδρία σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Θα διακόψουμε τώρα και στις 3 η ώρα θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας με μια ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Αναπληρώτη Πρωθυπουργέ και θα τα ξαναπούμε στις 3.